Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε και πάλι τις εργασίες μας για σήμερα το απόγευμα για να μην χάνουμε χρόνο και αναγκαστούμε να κρατήσουμε τους διερμηνείς μας περισσότερο από όσο χρειάζεται, λέει η Πρόεδρος. Ερχόμαστε στη συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την έκθεση του κυρίου Κόζα. Πρόκειται για κοινέ διατάξεις για τα ευρωπαϊκά ταμεία και κατάργηση του κανονισμού 1083 του 2006. Πρόκειται για το περίφημο CPR, όπως το λέμε συνοπτικά. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι θέλω να σας παρουσιάσω κάπως πώς έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε, συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο με την ε, Επιτροπή την Περιφερειακή δηλαδή, εδώ και εννέα μήνες. Κάθε εβδομάδα συναντιόμαστε για να δουλέψουμε πάνω στην πρόταση κανονισμού αυτού. Αποτελώ μέρος κι εγώ της διαπραγματευτικής ομάδας, διότι χάρη στον κανονισμό και χάρη στο άρθρο 81 του κανονισμού μας, η δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Είναι μέρος δηλαδή των διαπραγματευτών. πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιάστηκε η τελική έκθεση. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε, πιστεύω, να καταλήξουμε και σε τελική συμφωνία. Παραμένουν όμως κάποια σημεία στη συμφωνία αυτή που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Οι διαπραγματεύσεις ήταν περίπλοκες και κράτησαν πάρα πολύ. Έκανα τα πάντα προκειμένου να παρουσιάσω τις δικές μας απόψεις και να προστατεύσω τα δικά μας συμφέροντα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών. Πριν μπω στις λεπτομέρειες, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω τα εξή στοιχεία. Όσον αφορά την εντολή. Είναι η εντολή της Περιφερειακής Επιτροπής, της Επιτροπής Ρέγγι. Εγώ όμως έπρεπε να σεβαστώ την εντολή αυτή, εκτός εάν χάρη στην επιμερισμένη αρμοδιότητα μπορούσα και εγώ να διατυπώσω τις δικές μας απόψεις. Με δύο λόγια, θα σας παρουσιάσω τώρα ποιες είναι οι δικές μας οι θέσεις. Ένας από τους στόχους μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν να μιλήσω για μια όσο γίνεται πιο απλή διαδικασία προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. 130 σελίδες πλημμυριστήκαμε. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές διατάξεις. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρξει μια απλοποίηση που όμως δεν πέτυχε τελικά. Παραμένουν 130 σελίδες. Είναι σημαντικό για μας η διαδικασία αυτή να είναι πιο απλή και πιο σαφής. Οι κανόνες για τις πληρωμές έχουν γίνει πάρα πολύ περίπλοκοι. Και ακριβώς γι' αυτό και η διαδικασία έχει γίνει περίπλοκη και άκαμπτη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από συμβάσεις εταιρικής σχέσης προβλέπει τρεις μήνες αρχικά. Ο συμβιβασμός μιλάει για τέσσερις μήνες. Να ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Όσον αφορά τους δικαιούχους των ταμείων αυτών. Θα θέλαμε η διαδικασία να απλοποιηθεί για τους δικαιούχους και η Επιτροπή ΡΕΓΚΙ, η Περιφερειακή Επιτροπή, συμφωνεί μαζί μας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν η εισαγωγή και η συνεργασία με τους εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για το άρθρο 5 που αφιερώνεται σε αυτό το θέμα. Έπρεπε επίσης να διευκρινιστεί και το θέμα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο έγινε. Έρχομαι τώρα στην επιφύλαξη της αποδοτικότητας για 5%. Αυτό βγήκε. Εμείς θέλαμε και η πρόταση αυτή 5% διορθώνει ο μιλητής, θέλαμε να βγει, αλλά δεν τα καταφέραμε τελικά. Τώρα θα συνταχθεί μια έκθεση το 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναφέρεται στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Αυτά ήταν λοιπόν τα στοιχεία τα οποία μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση της Ρέγγι. Θέλω όμως να αναφερθώ και σε τρία άλλα ζητήματα. Πρώτον, τοπική στρατηγική. Υπάρχει η τοπική πτυχή και η εταιρική σχέση. Καταφέραμε να καταλήξουμε στο 45% για τη συμμετοχή αυτή και χάρη στο 45% οι κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού θα τηρηθούν. Ένα άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την αγορά γεών. Ήταν κάτι που έλειπε κάπως από τον κανονισμό αυτόν. Ενώ τώρα μιλάμε για την αγορά γεών με τα κονδύλια αυτά. Τέλος. Θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Με την πρόεδρο έχουμε ανταλλάξει απόψεις. Πρόκειται για το άρθρο 84. Πρόκειται για τα ελάχιστα ποσά του κοινωνικού ταμείου. Εμείς λέγαμε 25% και ένα ευέλικτο πλαίσιο. Μετά θα έχουμε και την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που επίσης αναφέρει την επιθυμία μας αυτή για 25%. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας και στον τριμερή διάλογο θέλαμε να το πετύχουμε το ποσοστό αυτό. Τα πράγματα βέβαια μετά άρχισαν πιο γρήγορα. Στην αρχή είχε προσπαθήσει για το ελάχιστο ποσοστό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το Συμβούλιο ήθελε να μπλοκάρει τα πράγματα. Τώρα θέλουμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις. Πάντως φαίνεται ότι τώρα και το Συμβούλιο θέλει να προχωρήσει και να έχει συζήτηση μαζί μας για να τουλάχιστον 25% των πόρων των διευθυντικών ταμείων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. χρειάζεται να διευκρινιστούν και κάποια τεχνικά ζητήματα. Πριν από κάποιες εβδομάδες υπήρξε μια συμβιβαστική πρόταση Η Επιτροπή μας συμφώνησε, ήταν παρούσα και η Πρόεδρος στην ανταλλαγή αυτή απόψεων. Τρεις υπέγραψαν μια επιστολή η πρόεδρος, η εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εγώ, οι τρεις μας δηλαδή που γράψαμε την επιστολή αυτή και τη στείλαμε στην Επιτροπή Ρέγγι, την Περιφερειακή Επιτροπή. Τώρα θα δούμε ποια λύση θα ακολουθήσουμε. Δεν είναι σαφές αν θα μιλάμε για το 25% στο κείμενο. Θα δούμε μήπως αντί για το 25% βρούμε κάποιες άλλες τεχνικές λύσεις για να καταλήξουμε στο ίδιο. Πάντως το Συμβούλιο κατάλαβε ότι το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό είναι έτοιμο τώρα να μας προτείνει μια συμβιβαστική λύση που να μπορούμε και εμείς να αποδεκτούμε. Είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Επειδή οι ομάδες ε, διαπραγματεύσεων ε, έχουν ε, κοινά σημεία, θα πρέπει να, το δούμε, να τα δούμε μαζί με το ΕΚΤ, δηλαδή το σημείο 14, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος ως Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ θα μας πει πού βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις με τον κανονισμό του ΕΚΤ. Πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χτες το βράδυ έγινε ο τελευταίος τριμερής διάλογος υπό ε, την Ιρλανδική Προεδρία. Δεν είναι τελευταίος στη σειρά γενικότερα. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε αυτή την ε, εργασία συντονισμού των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν ήταν εύκολο. Οι δύο τελευταίοι τριμερείς ε, διάλογοι αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις για τους δείκτες και μπορώ να σας πω λίγα λόγια για την εργασία μας ως προς τους δείκτες διότι ε, είδαμε ότι στην απογραφή των δείκτων δεν έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε κανέναν αρνητικό δείκτη που θα μπορούσε να ε, προβεί σε μετρήσεις ε, δυσχερίων ή δυσκολίων γενικότερα, αλλά μόνο θετικά στοιχεία και στη συνέχεια επαγωγικά θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε ορισμένα προβλήματα που αφορούν το ΕΚΤ. Η δεύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στα πλαίσια αυτών των εργασιών για τους δείκτες ε, έχει ως εξής. Η... Ό,τι αφορούσε τη σχέση μεταξύ ACT και Youth Employment Initiative. Είδαμε ότι στα πλαίσια του ACT έχουμε αυτή την εγγύηση για τους νέους αλλά η σχέση μεταξύ του, της πρωτοβουλίας απασχόλησης των νέων και τα Εγγύησης για των νέων δεν είναι σαφής. Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων αποτελεί ένα ε, πολιτικό καθαρά δείκτη, ενώ εμείς θέλουμε δίκτες που να μπορούν να μετρήσουν έμπρακτα αυτή την πολιτική. ενώ είναι ιδιαίτερα σαφείς οι δείκτες που έχουμε επί του θέματος. Νομίζω ότι από τους ε, δύο τελευταίους ε, τριμερείς ε, διαλόγους μπορούμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι γνωμοδοτήσαμε για το σύνολο των δικτών, αλλά έχουμε πολλά να κάνουμε με την Λιθουανική Προεδρία και προτείναμε όχι διαπραγματεύσεις, αλλά επαφές με τη νέα Προεδρία, είτε στο Στρασβούργο στις 4 Ιουλίου, είτε στις Βρυξέλλες στις 10. Όσον αφορά τις ε, συνολικές διαπραγματεύσεις για το minimum share του act θα ήθελα να πω τα εξής là encore une grosse... Euh, Αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες στη διαπραγμάτευση. Ο συνάδελφος Κώσα μας είπε ότι όλοι θέλουμε το 25% αλλά στις διαπραγματεύσεις αυτό το 25% αμφισβητείται σοβαρά από πλευρά Συμβουλίου. Δηλαδή το Συμβούλιο βρίσκεται πολύ μακριά. Ήδη και ως Κοινοβούλιο δεν συμφωνούμε επί της ποσοστιαίας αυτής αναλογίας και όφιλα να το υπενθυμίσω. Οι τεχνικές λύσεις που έδειξε ο Άνταμ Κόσα δεν μας ικανοποιούν γιατί για να φτάσουμε σε αυτό το 25% αυτή, αυτή, αυτό το ελάχιστο μερίδιο, το minimum share, έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθεί και το ΕΤΠΑ, γιατί μας ενδιαφέρουν και οι κοινωνικές διευκολύνσεις για να φτάσουμε σε αυτό το 25%. Δηλαδή, τώρα είμαστε ε, γνώστες του ΕΚΤ, στρίκτο σένσου, αλλά ως προς το ΕΤΠΑ δεν, δεν γνωρίζουμε το ζήτημα πώς εξελίσσεται για να φτάσουμε στο 25%. Δεν ξέρω κατά πόσο μας ικανοποιεί, εμένα τουλάχιστον όχι εάν λάβουμε υπόψη την εντολή που μας έχει ανατεθεί και που ήταν σαφής. Ε, παράλληλα, από το 89 είδαμε την εξέλιξη του ΕΚΤ σε σχέση με το ΕΤΠΑ. Και βλέπω και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό στην περίοδο 89-93 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εκπροσωπούσε, αποτελούσε το 40% του ΕΤΠΑ αλλά το 7-13 μόνο το 25%, 28% συγχωρείτε. Αν λάβουμε υπόψη και την κρίση που αντιμετωπίσαμε, από το 2008 και μετά και με τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε επίπεδο κοινωνικής σύνοχης δεν μπορούμε να αρκεστούμε. σε αυτή την συμπλήρωση του ΕΚΤ από την ΕΤΠΑ σε αυτό το συμπλήρωμα που θα δινόταν από το ΕΤΠΑ. Γιατί αυτό δεν ε, τάσεται υπέρ της κοινωνικής συνοχής. Και εμείς προβλέπουμε λύσεις στην ομάδα διαπραγμάτευσης και ιδιαίτερα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο ΕΚΤ έχουμε αναλάβει και την επισητιστική βοήθεια για τους πλέον φτωχούς, 3 500, εκατομμύρια και γι' αυτό θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη συμπληρωματικά και το ίδιο αφορά και το Ταμείο ε, Συνοχής. Υπάρχει η πολιτική συνδέοντα στην Ευρώπη, την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για να υπολογίσουμε τις νέες ποσοστιαίες αναλογίες για την κοινωνική συνοχή. Αυτά εντάχει, κυρία Πρόεδρε, ως προς την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Βλέπετε και τα περιθώριά μας. Θα ήθελα να πω σε όλα τα μέλη όλων των πολιτικών ομάδων ότι μας έδωσαν, μας ανέφεσαν μια σαφή εντολή. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ δύσκολες ε, έναντι του Συμβουλίου και οι διαπραγματεύσεις υπό Ιρλανδική Προεδρία δεν ήταν καθόλου εύκολες, αλλά οπωσδήποτε θα κινήσουμε και τα επιπρόσθετα αυτά ζητήματα τα οποία σας ανέφερα. Ποιοι θα ήθελαν το λόγο στη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Γκουτιέρ. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για τις ε, πληροφορίες, για την εξέλιξη των ε, διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαπραγμάτευση για τα δύο αυτά τα ζητήματα που είναι ύψης της ε, σημασίας για την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και τη συνάδελφο και τον κύριο Κώσα, διότι ε, μιλάμε για μία μεγάλη διαπραγμάτευση μέσα στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή Ρέτζη, διότι το άρθρο 84 του ΕΚΤΑ αναφέρεται σε ένα 25% που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εμείς το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές σε πολλές εκθέσεις, σε ψηφίσματα, στην Ολομέλεια και ε, κερδίσαμε, το προωθήσαμε δηλαδή. Δεν πρόκειται για διελκυστίνδα ε, Επιτροπής Απασχόλησης έναντι Ρέτζι. Είναι ε, συνολικό ζήτημα, θέμα που προωθούμε από κοινού. Βεβαίως έχουμε χάσει ως ΕΚΤ έναντι των Ταμείων Συνοχής διότι η θεματολογία μας είναι η απασχόληση, ο κοινωνικός αποκλισμός και η καταπολέμηση της φτώχειας μέσα στα πλαίσια της ΕΚΤ. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε κονδύλια κατά τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Όπως είπε η κυρία Σάρτχε, τα νέα μέσα που διαθέτει το ΕΚΤ, δηλαδή η εγγύηση υπέρ των νέων και το Ταμείο Βοήθειας για τους Απόρους. Μιλάμε για 6 ε, εκατομμύρια λιγότερα, ιδιαίτερα στα πλαίσια του ΕΚΤ. Θα ήθελα λοιπόν, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, να ε, ζητήσω να προωθήσουμε αυτή τη νομιμότητα του ζητήματος εξ ονόματος ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύο άλλα θέματα. Πώς έχει η διαπραγμάτευση στους ε, ε, τριμερείς διαλόγους ως προς την μεταβιβασιμότητα μεταξύ ταμείων, γιατί και αυτό ε, θα αποτελούσε ε, δύο διαφυγής σε ορισμένες περιπτώσεις. Εκεί όπου δεν υπάρχουν περιθώρια λιγμού για τις επενδύσεις, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα ε, μεταβίβασης κονδυλίων μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Πώς έχει και το αποθεματικό του ΕΚΤ του 20% για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Γιατί έμαθα ότι αυτή ποσοστία αναλογία αμφισβητείται ή συζητείται στους τριμερείς διαλόγους. Αυτές ε, είναι οι ερωτήσεις μου και θα ήθελα ορισμένες ε, αποσαφηνήσεις ή δυνατόν. Ευχαριστώ. Άλλοι που ζητούν το λόγο. Όχι. συνδέοντας τα δύο ζητήματα, δηλαδή το θέμα του άρθρου 84 ε, σημείο 3 του κανονισμού ΣΕΠΕΡ και των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ε, υπέρ του ΕΚΤ. Στη διαπραγμάτευση αυτή, αυτό που απασχόλησε αποτελεί θέμα γενικότερα ε, γιατί το 20% για την καταπολέμηση της φτώχειας και τον κοινωνικό, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ε, συμπεριλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις. Ξέρετε ότι έχουμε ε, μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις εάν δεν προϋπάρξει συμφωνία ως προς το αντίστοιχο τμήμα του κανονισμού ΣΕΠΕΡ Δηλαδή, αν δεν συμφωνήσουμε για το 25% του ΕΚΤ, για τα χρήματα της πολιτικής συνοχής, δεν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Όμως η ομάδα διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Απασχόλησης όταν έπρεπε να δεχτεί και όταν μιλήσαμε για μείωση σε 23,5% για το ΕΚΤ, εμείς είπαμε ότι για μας ε, ήταν ένας από τους απαράβατους όρους ε, της ε, διαπραγμάτευσης πέρα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Το Συμβούλιο είπε ότι ε, πας περιπτώσει δεν το συζητάμε. Εμείς όμως δεν συμφωνούμε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα γίνει η κατανομή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι το 20% που αφορά τη φτώχεια και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολύ σημαντικό. θα ήθελα να σας πω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα σε αυτή την διαπραγμάτευση. Υπάρχει πίεση για λήξη των ε, διαπραγματεύσεων, διότι λύγει και η Ιρλανδική Προεδρία και οι τοπικές αρχές ε, πιέζουν. Χάσαμε ένα χρόνο περίπου πριν γιατί δεν είχαμε ε, τη νομική βάση για να, διοργανώσουμε, για να οργανώσουμε τους διαγωνισμούς και τα λειτουργικά προγράμματα, διότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα φορτωμένη διαδικασία. Υπάρχει μεγάλη πίεση λοιπόν, ακόμα και από συναδέλφους της Περιφερειακής Επιτροπής να ολοκληρώσουμε. Επειδή όμως ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε πλήρως το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να αντισταθούμε κατά τις ε, διαπραγματεύσεις του Φλεβάρη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το μερίδιο του ΕΚΤ ήταν ικανοποιητικό, δηλαδή μιλούσαμε για ένα ποσοστό της τάξης του 25%. Τώρα, στην τελευταία ευθεία των διαπραγματεύσεων, βλέπετε στο κάτω μέρος της σελίδας μία υποσημείωση ή μία μικρή προσθήκη μέσα στα πλαίσια της νέας θέσης του Συμβουλίου και όταν αποκωδικοποιήσετε βλέπετε ότι έχουν μπει πολλοί λύκοι στη στάνη μας για να μειωθεί η βάση υπολογισμού του 25%. Δηλαδή η τελευταία θέση του Συμβουλίου που δεν μας έχει διαβιβαστεί επίσημα, αλλά που ανακαλύψαμε αναφέρεται στο ότι υπολογίζουμε το 25% επί του ΕΚΤ πλην του συνδέοντα στην Ευρώπη, εκτός δηλαδή του Connecting Europe. Άρα μειώνεται αυτό το 25% του ΕΚΤ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από την Περιφερειακή Επιτροπή και την ε, Ιρλανδική Προεδρία για να ολοκληρώσουμε αύριο στις 8. Νομίζω ότι τα περιθώρια διαπραγματεύσεων μας είναι πολύ χαμηλά. Μιλάμε για ένα 23,5% το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε είτε πρόκειται για ευρεία βάση, είτε πιο, την πιο συσταλτική ερμηνεία, χωρίς το Connecting Europe και χωρίς το Ταμείο Βοήθειας τους, ε, πλέον για τους απόρους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να δούμε αν το ταμείο για τους απόρους είναι εντός ή εκτός, μάλλον είναι εκτός. Και από πολιτικής πλευράς νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια στεναρή στάση πέρα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου. Βλέπω ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, του Συμβουλίου. Τις διαβλέπω από το Φεβρουάριο και μετά καθώς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανακοίνωση για την κοινωνική πτυχή για την ΟΝΕ, μίλησαν για την απασχόληση των νέων. Να, και άλλο νέο στοιχείο που ανέκυψε και το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου δίνει βαρύνουσα σημασία στο ΕΚΤ και σε πάνω από ένα κεφάλαιο. Γιατί μιλάει για την απασχόληση των νέων. Αναφέρεται στην απασχόληση των νέων και στο μέσον για την κινητικότητα των νέων. ανοιχνεύουν ό,τι μπορούν δηλαδή για να προωθήσουν κοινωνικές πολιτικές υπέρ της απασχόλησης και ιδιαίτερα της απασχόλησης των νέων που μας αναπέμπουν στο ΕΚΤ. Έχουμε όλα λοιπόν τα στοιχεία στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Ο καθένας βεβαίως θα αναλάβει τις ευθύνες του. Γνωρίζετε ότι το θέμα αυτό στο θέμα αυτό θα πρέπει να αποφανθεί το Συμβούλιο που θα παίξει το ρόλο του διαιτητή. δεν αφορά γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής γιατί στο Διευθυντήριο και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης βλέπουμε ότι την χάνει της υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης για την Περιφερειακή Πολιτική. Θα δούμε αύριο προβλέπεται μία ώρα διαπραγματεύσεων. Δεν είναι πολύ. Θα, θα δούμε. Δεν θα, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε ότι θα μας κατηγορήσουν ότι μπλοκάρουμε τις διαπραγματεύσεις, διότι το πολιτικό διακύβευμα είναι πολύ υψηλό. Κατά τα άλλα όλα ακολουθούν την πορεία τους. Απομένει ένα σημείο που θα πρέπει να δούμε μαζί πώς θα προσαρμόσουμε την μέθοδο εργασίας με βάση την έκθεση Άνταμ Κόζα, δηλαδή την, την Περιφερειακή Επιτροπή. Θα θυμόσαστε ότι η Περιφερειακή Επιτροπή είχε ε, φτάσει σε μία καινοτόμο πρόταση, η διαδικασία, πρωτότυπη τουλάχιστον, δηλαδή πέρσι στις 5 Ιουλίου ενέκρινε το σχέδιο γνωμοδότησης του Άνταμ Κόσα, αλλά δεν ψηφίσαμε παρά τις τροπολογίες για να βασιστούμε στην ε, πρόταση, στη μεθοδολογία της Ρέτζη. Γιατί ήθελε να γίνουν διαπραγματεύσεις μόνο βάσει τροπολογιών και όχι ε, βάσει της τελικής ε, γνωμοδότησης, δυνάμει του άρθρου 70 και ούτω καθεξής δεν ετέθη ε, θέμα ε, εντολής διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, η Περιφερειακή Επιτροπή επινόησε αυτή την πρωτότυπη διαδικασία για να εισαγάγει μία προθεσμία τροπολογιών ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Άρα η, Επιτροπή, η Περιφερειακή Επιτροπή έχει θέσει προθεσμία για την έκθεση Βανίστελ Ρόι και Κωνσταντσε Κρέλ. Θα ψηφίσουν λοιπόν αυτή την ε, ε, έκθεση. στις 11 Ιουλίου. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να αρκεστούμε σε αυτή τη διαδικασία, να προσαρμοστούμε. Συζητήθηκε το θέμα στους συντονιστές για να δούμε πώς θα το επιτύχουμε για τις κοινέ διατάξεις για τα ευρωπαϊκά ταμεία και επειδή υπάρχει κοινή συνεργασία επιτροπών δυνάμει του άρθρου 81 του κανονισμού θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να στοχοθετήσουμε την παρέμβασή μας για να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και να ορίσουμε μια νέα προθεσμία υποβολής τροπολογιών για την έκθεση Κόσα. δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 3 αποκλειστικά. Στην αρχική έκθεση Κόσα και στο θέμα που προσθέσαμε πέρσι τον Απρίλιο σε σχέση με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Υπ' αυτή την έννοια, εάν συμφωνείτε, θα ορίσουμε προθεσμία υποβολής τροπολογιών για τις 26 Ιουνίου, δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 3, θα το συζητήσουμε στις ε, 8 Ιουλίου και θα ψηφίσουμε στις 11. Δύο μέρες πριν αποφανθεί η Περιφερειακή Επιτροπή. για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών, για να έχουμε την ίδια προσέγγιση όπως είχαμε και για την έκθεση Κόσα. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Ελπίζω να ήμουν σαφής sur ce point. Non, Αλλά θα ήθελα να σας δώσω το λόγο ε, πριν ε, καταλήξουμε ως προς αυτό το σημείο. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στη διαδικασία Ρέτζι, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε επί του βασικού σημείου των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή το μερίδιο του ΕΚΤ μέσα στα πλαίσια των Ταμείων Συνοχής. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στους δύο εισηγητές, εάν θέλουν. Ο Άνταμ Κόσα θέλει να ξαναλάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας, καθώς και και την πρόεδρο που συνοψίσατε τα πράγματα. Εμείς εξετάσαμε το πρόβλημα από όλες τις πτυχές και νομίζω ότι αύριο που γίνεται έκτακτη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου διάρκειας μιας ώρας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα αποτελέσει τον στόχο όλης της προσοχής μας. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν το Συμβούλιο πρόκειται να υποβάλει νέα πρωτοβουλία. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει τη δική μας στάση. Είναι σημαντικό να περιλάβουμε το κείμενο στη γνωμοδότησή μας και να μπορέσει να εγκριθεί στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και σε την 26η Ιουνίου που είναι προθεσμία καταθέσεως των απολογιών νομίζω ότι πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες παρόμοιες με αυτές που έχουμε ήδη καταθέσει γιατί η στάση μας πρέπει να είναι ενωμένη. Η κυρία Σάτιε, ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι το τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως είπε το Συμβούλιο, που έχει υποτίθει ικανοποιητικό χαρακτήρα, δεν σημαίνει αυτό το ικανοποιητικό το ίδιο για το Συμβούλιο όπως για μας. Αν λοιπόν μπορώ να συνοψίσω την θέση της διαπραγματευτικής ομάδος, το ικανοποιητικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής για το 2014 έως 20 είναι 23,5% των πόρων της συνοχής μέσα σε αυτά και η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη Ε, τα 23 λοιπόν 5,5%. Και αυτή τη γραμμή θα υπερασπιστούμε αύριο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εγγύηση ε, νέων, υπέρ των νέων, την πολιτική για τους νέους, την βοήθεια για τους ε, πλέον απόρους και ούτω καθεξής. Ένα τμήμα ικανοποιητικό για την Επιτροπή Απασχολήσεως. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι για το 13 την έκθεση του κυρίου Κοζά ανοίγουμε ξανά την προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών μόνο για το 83 στα αγγλικά και για τις 26 έκτου. Θα ψηφίσουμε στις 9 Ιουλίου μετά από διεξαγωγή συζητήσεων θα γίνει στις 8. Συζήτηση 8, ψηφοφορία 9. Έχουμε τώρα το 15 και θα δώσω το λόγο στον Αλεχάνδρο Σέρκας για να μας εξηγήσει τα της αποστολής αυτής. Α, δεν είναι εδώ. Κρίμα. Τότε λοιπόν θα προχωρήσω μέσω στο 16 και δίνω το λόγο στην κυρία Εσαγιά για να παρουσιάσει το σχέδιό της, σχέδιο εκθέσεως δηλαδή, για την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που τροποποιεί έναν αριθμό οδηγιών έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό 1272 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Κυρία Ισηγήτρια. Α, μόλις ήρθε ο κύριος Σέρκας, κυρία Πρόεδρε. Συνεχίζω παρά τα αυτά. Καλώς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κανονισμός λοιπόν 1272 του 2008 για ταξινόμηση, επισήμαση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ευθυγραμμίζει την φυστάμενη κοινοτική νομοθεσία με το σύστημα των ΗΕ Εθνών G8S σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση επικίνδυνων χημικών ουσιών και ενημέρωση για τους κινδύνους των χρηστών σε επισήμανση, ετικέτες δηλαδή και συνοδευτικά φυλάδια. Μετά από την υιοθέτηση του σχετικού κανονισμού προέκυψε η ανάγκη τεχνικής ευθυγράμμισης με τις οδηγίες αυτές που εξήγησε ήδη η Πρόεδρος που περιλαμβάνουν παραπομπές στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ταξινόμησης. Η σχετική δε ορολογία των πέντε οδηγιών οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό CLB που ωστόσο δεν καθιστά αναγκαίες αλλαγές στο πεδίο εφαρμογή των οδηγιών αυτών. Ούτε θεωρώ άλλωστε χρήσιμο να μπούμε σε τέτοια διαδικασία τουλάχιστον στο παρόν χρονικό σημείο. Γι' αυτό οι τροπολογίες για τις πέντε οδηγίες που προτείνει η Κομισιόν είναι καθαρά τεχνικές όπως άλλωστε και αυτές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο εκθέσεως. Όμως είναι σαφές ότι και οι πέντε οδηγίες πρέπει να ανανεωθούν το δυνατόν συντομότερο έτσι ώστε να είναι συνεκτική η νομοθεσία και επαρκής η προστασία απέναντι σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται σε τόπους εργασίας. Εγώ έχω διαβιβάσει και σχετικό σημείωμα στην αιτιολογική σκέψη. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αναμειχθούμε υπερβολικά στα καθαρά τεχνικά θέματα, τα οποία δεν απαιτούν λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ωστόσο προσπάθησα να κάνω τις απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις, εκεί όπου δηλαδή σημείωσα ελλείψεις στο κείμενο της Κομισιόν τουλάχιστον, όπως το ερμηνεύω εγώ. Και έχω περιλάβει και αιτιολογήσεις των τροπολογιών μου, ίσως δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω τώρα, το βασικό θέμα είναι να προσαρμοστούν οι οδηγίες στην ορολογία και ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων του κανονισμού με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο. Οι μεγαλύτερες αλλαγές έγιναν στο άρθρο 1 για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασία. Όλα τα δοχεία τα οποία απαιτούν ε, σχετική επισήμαση πρέπει να περιληφθούν εδώ. Έχω βάλει επίσης και το υπόλοιπο του άθου 1 που ε, κατά παράβλεψη το είχε ε, διαγράψει η Κομισιόν. Η 1η Ιουνίου του 2015 είναι σωστό να αρχίσει η εφαρμογή της οδηγίας, διότι είναι και η βασική ημερομηνία που αναφέρει ο κανονισμός για την ταξινόμηση των μειγμάτων. ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των μειγμάτων ο, σύμφωνα και με τον 1.99, με τον 19 μάλλον, 99, 45. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν θα δούμε αν θα διατυπωθεί σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, αλλά όταν τέθηκε το θέμα αυτό, εγώ προτίμησα να το αφήσω καλύτερα για όταν θα αναδιατυπωθούν σε βάθος οι πέντε οδηγίες. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας λέμε ότι κάποιες νομοθετικές πράξεις είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. Όταν όμως αρχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτές, φαίνεται τελικά ότι έχουν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ωστόσο τολμώ να πω ότι σε τούτη εδώ την περίπτωση το θέμα είναι καθαρά τεχνικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, ο οποίος έχει και ε, μηχανολογική παιδεία και χωρίς τη βοήθειά του δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Όπως είπα, το θέμα είναι καθαρά τεχνικό. Θα ήθελα να ακούσω οι σκιώδεις συζητητές τι άραγε έχουν να σχολιάσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, μα είναι εδώ οι σκιώδεις. Όλοι Κρίστενσεν είναι παρόν. Του δίνω μέσω το λόγο. Άλλος κανείς επιθυμεί να εγγραφεί. Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, καθώς επίσης ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έργο που επετέλεσε έως τώρα. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασία είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για μας, εμείς στην σοσιαλιστική ομάδα ενώ αλλά βεβαίως και για το έργο συνολικότερο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το άρθρο 31, παράγραφος 1 του χάρτη λέει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εργάζονται σε περιβάλλον που προστατεύει την υγεία και την ασφάλειά τους. Η Κομισιόν λέει ότι θέλει να μειώσει κατά 25% τα εργατικά ατυχήματα και μάλιστα και μέχρι το 2010 και αυτό οφείλει να το τηρήσει. Η Κομισιόν έχει βάλει ερωτηματικά δίπλα σε ορισμένες από τις ρήτρες προστασίας των εργαζόμενων. Και αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, όπου υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Μετά μας είπαν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν υπερβολικά από άποψη γραφειοκρατική. Αλλά αυτά εδώ δεν μπορούν να θεωρηθούν γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Ο τεχνικός τίτλος της οδηγίας μόλις καλύπτει το γεγονός ότι στην πραγματικότητα πρόκειται εδώ για βελτίωση των συνθήκων εργασίας, διότι υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που πολύ συχνά μάλιστα τις χειρίζονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χειρίζονται μάλιστα και πολύ επικίνδυνα χημικά στις εργασίες τους. Δεν επιτρέπεται να λησμονούμε την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και να δούμε το θέμα καθαρά τεχνικά. Εγώ θεωρώ καλό ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τεχνολογική πρόοδος και πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και μια νέα τεχνολογική αξιολόγηση. Εμείς στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα φροντίσουμε ώστε να μην παραβλέψουμε οποιαδήποτε τεχνολογική πρόοδο και να πράξουμε πάντα δυνατό για την προστασία των εργαζόμενων. Ευχαριστώ για το σχέδιό σας και αναμένουμε ευχαρίστως τις περαιτέρω διαβουλεύσεις. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς? Καλώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε. Η κυρία Μωτίνου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στην πρόταση αυτή για οδηγία. Όπως είπε και η συγγήτρια, πρόκειται για ευθυγράμμιση πέντε οδηγιών στο νέο σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας ουσιών και μειγμάτων, παρασκευασμάτων. Θέλω να υπενθυμίσω ποιες ήταν οι εξελίξεις στο κανονισμό CPR για να οδηγηθούμε σε ένα ενιαίο σύστημα. Ξεκινήσαμε από δύο διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης και σήμανσης επακίνδυνες ουσίες και επικίνδυνα παρασκευάσματα. Οι πέντε οδηγίες δεν αναφέρονται σε δεύτερο πυλώνα απαιτήσεων σήμανσης ή σε νομοθεσία για την μεταφορά. Τώρα όμως εμπίπτουν και αυτά στα πλαίσια του κανονισμού CPR. Όταν ε, ετοιμάζαμε την πρόταση, την πρόταση οδηγίας, περιφήκαμε αντιμέτωποι με το ζήτημα ότι υπήρχε κάποιο συσχετισμό ανάμεσα στο προηγούμενο σύστημα και τον κανονισμό CPR, που όμως δεν είναι πάντα απευθείας. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο συσχετισμού για τις ουσίες και τα μείγματα που είχαμε από το παλιό σύστημα, ενώ συγχρόνως προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την συνέχεια και τον υψηλό βαθμό προστασίας. Όσον αφορά τις τροπολογίες που προτείνονται, βλέπουμε ότι Ανταποκρίνεται καλύτερα η τροπολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό ΣΕΡΠΗ. Αυτό ισχύει για τις τροπολογίες 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 και 17. Υπάρχουν άλλες που προσθέτουν κατηγορίες ουσιών και μειγμάτων. Αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμφωνούν και με τόσο αναφέρει η τροπολογία 1, η οποία θέλει να διασφαλίσει ότι η οδηγία θα παραμείνει προς αναθεώρηση ώστε να γίνονται ό,τι προσαρμογές χρειάζονται προς τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Θέλω τώρα να αναφερθώ, επιτρέψτε μου, στην τροπολογία 4. Η πρόταση της Επιτροπής συμπεριλαμβάνει την διατύπωση, την αρχική που είχαμε, τις οδηγίες του 2005, τον όρο labeled. Σήμανση. Ο όρος ταξινόμηση που προτείνεται στην τροπολογία 4, δηλαδή οι χημικοί παράγοντες που ταξινομούνται, αυτό αποτελεί αλλαγή, ενώ πριν αναφερόταν επισημένονται. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όλα αυτά που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα κοιτάξουμε καλύτερα. Κυρίως γιατί όπως είπα δεν θα κάνουμε αλλαγές στην ουσία της οδηγίας. Θέλουμε απλώς να διέπεται από συνοχή η νομοθεσία μας. Και ο κανονισμός αυτός να κάνει αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Οπότε ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και ευχαριστώ και τον μοναδικό σκιώδη που έχω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών 27 Ιουνίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 26 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας. Και έτσι πάμε τώρα λίγο πίσω και πάμε στο σημείο 15 που είναι η αποστολή αντιπροσωπείας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Βίλνιου στην Λιθουανία. 2 και 3 Μαΐου. Την παρουσίαση θα μας την κάνει ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας, ο Αλεχάνδρο Θέρκας. Ίσως μετά, αν κάποιος άλλος θέλει, Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας όμως, πρώτο, ο κύριος Θέρκας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα, όπως είπατε και εσείς, 2 και 3 Μαΐου πήγαμε στο Βίλνιους. Ήταν μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ήταν η κυρία Τζιν Λάμπερτ, η Λιθουανή συναδελφός μας, ο Αλιτσούτε, και εγώ ίδιος που πρόεδρευα της αντιπροσωπείας. Όπως συμβαίνει συνήθως, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, εξωτερικών, με κοινωνικούς εταίρους, με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επισκεφτήκαμε διάφορα προγράμματα των διευθυντικών ταμείων, αλλά κάναμε και κάποια καινοτόμα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας υποδέχτηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και συναντηθήκαμε και με μια οργάνωση για την ισότητα των δύο φύλων. Από τις επαφές που είχαμε με την κυβέρνηση, στόχος ήταν να δούμε λίγο τι θα γίνει στην Προεδρία τη Λιθουανική που 1 1η Ιουλίου και να δούμε και πώς έχει κοινωνική κατάσταση στη χώρα αυτά αυτή. Εξετάσαμε διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν τακτικά. Σε όλα όσα συζητήσαμε για τα κονδύλια, για την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους κτλ. Η Προεδρία της Λιθουανίας ήταν καλά προετοιμασμένη. Βέβαια υπάρχει κάποια ανασφάλεια γιατί είναι η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά που μια βαλτική χώρα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ατζέντα τόσο περίπλοκη. Υπάρχει και κάτι χαρακτηριστικό. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, μίλησε για τα οικονομικά, την κρίση κτλ. Η πρόεδρος είναι πολύ γνωστή και μπήκε σε ζητήματα πολιτικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μερικές φορές ήταν δύσκολη η συζήτηση γιατί η θέση της ήταν αρκετά σκληρή όταν εμείς κάναμε παρατηρήσεις για το Συμβούλιο και λέγαμε ότι είναι άκαμπτο. Εκείνη αμέσως άλλαζε και έκανε άλλου είδους επιθέσεις για το τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποια στιγμή έθεσε υπό αμφισβήτηση την αντιπροσωπευτικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλιστα έδειχνε να μην γνωρίζει ότι δύο νομοθέτες είναι επίση όρις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εάν η πρόεδρος δεν, αντιλαμβάνεται ότι έχουν περάσει κυρία εκείνη που υπήρχε ένας και μόνο επικεφαλής και όλοι τον ακούγανε, ε, αυτό θα είναι πρόβλημα. Πήγαμε όπως σας είπα και στο Ινστιτούτο για την ισότητα των δύο φύλων. Εκεί Υπάρχουν διάφοροι εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες, οι οποίοι κάνουν έρευνες, τις οποίες και κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη θέση της γυναίκας και για την ισότητα των δύο φίλων. Μας μίλησαν για μια μελέτη που κάνουν για τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή και επικεντρώνονται στη μελέτη τους αυτή πάρα πολύ καλά στο ζήτημα των αδειών πατρότητας που μόνο στην Δανία και στη Σουηδία υπάρχουν. Είναι δηλαδή λίγο πολύ αυτά τα οποία εμείς ζητάμε ότι πρέπει να είναι εξίσου υπεύθυνοι άντρες και γυναίκες για την οικογενειακή ζωή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η επίσκεψη και νομίζω ότι η μελέτη αυτή θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να ξέρουμε πώς προχωράμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τις επαφές μας. Η Λιθουανική Προεδρία θα κάνει σίγουρα κάποια προσπάθεια, παρόλο που ξέρουν ότι στην ταυρομαχία αυτή ο Ταύρος θα είναι δύσκολος. Είναι όμως διατεθειμένοι να προσπαθήσουν και νομίζω ότι θα ασχοληθούν και με πολλά από τα πράγματα που μας απασχολούν και εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν κάποιοι από τους συνομιλητές σας το τι σημαίνει δύο συνομοθέτες, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι δεν θα είναι με αυτούς που θα πρέπει να διαπραγματευτεί το Κοινοβούλιο. Την πρώτη δοκιμή την είχαμε με την Ιρλανδική Προεδρία. Γιατί όπως είπε και η συγκεντριά μας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Στρασβούργο θα συναντηθούμε μετά για μια πρώτη επαφή. Η Υπουργό θα έρθει στην Επιτροπή μας, σωστά, στις 9 Ιουλίου. 12 Ιουλίου εγώ θα πάω στη Λιθουανία για να συμμετάσχω εκεί σε ένα τύπο συμβουλίο. Οπότε θα επαληθεύσουμε αυτά τα οποία εσείς μας παρουσιάσατε μόλις τώρα. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τώρα είναι το σημείο 17. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης που πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας για την οικοκαινοτομία. Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η συγητής είναι ο κύριος Φιλ Μπενιόν. Έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, προβάλλει μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, για να δημιουργήσει απασχόληση και ανάπτυξη για την οικοκαινοτομία. Εμείς συμβάλλουμε γιατί υπάρχουν ε, νέες δυνατότητες απασχόλησης από την πολιτική οικοκαινοτομίας, ιδιαίτερα για το μέλλον, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα λοιπόν τομέων ε, στη βιοτεχνολογία που μπορεί να δημιουργήσει ε, νέες θέσεις εργασίας. Ελπίζω να ε, υποβάλλετε τροπολογίες σε αυτή τη σύντομη έκθεση και ελπίζω να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Εμείς έχουμε θέσει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο μέσω της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μέσα στα πλαίσια της Ένωσης Καινοτομίας για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα ε, πράσινη ε, επανάσταση για να προωθήσουμε τη βιώσιμη απασχολησιμότητα. Επίσης, οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να κρατήσουμε την ηγετική μας θέση σε αυτές τις τεχνολογίες και να μην ε, εισάγουμε αγαθά από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε η ε, επικεφαλής. Βεβαίως η οικονομική ε, κρίση έχει οδηγήσει σε πολιτικές λιτότητας όπου δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις. Γι' αυτό η επένδυση σε στρατηγικά προϊόντα θα είναι ύψη της σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας και τους περιφαλλοντικούς στόχους και την καινοτομία για καλύτερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές και την καλύτερη απασχόληση στους πράσινους τομείς όπως και επειδή επειδή εξυγχρονιζόμαστε θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τον βιομηχανικό τομέα και τον τριτογενή τομέα και να μιλήσουμε για νέους ε, τομείς. Η οικοκαινοτομία μπορεί να ε, οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας από την έρευνα και τεχνολογία καθώς ε, και ποικίλε άλλες ευκαιρίες. Αυτή η ε, διαφορετικότητα και ποικιλία θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να βρουν εργασία ανάλογα με τις δεξιότητές τους και τη δυνατότητα κατάρτισης για να μεταβούμε σε αυτά τα νέα πράσινα project. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για την περιβαλλοντική ε, ανάπτυξη, αλλά για να έχουμε βιώσιμη, βιώσιμες επενδύσεις μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Περιμένω την συνεισφορά των ε, συναδέλφων έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταρτήσουμε μια πολύ καλή έκθεση. George και μετά ο Αλεχάνδρο Θέρκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα για την γνωμοδότησή σας εξήγησε άλλωστε την κατάσταση σωστά. Ο εισηγητής τόνισε και τις σημαντικές προκλήσεις. Νομίζω η Κομισιόν έχει διατυπώσει καθαρά τους στόχους που οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς. Κυρίως καινοτομία που είναι και το όχημα της ανάπτυξης και βεβαίως η η οικολογική καινοτομία. Βεβαίως η έρευνα και οι σχετικές επενδύσεις. Για μας σημαντικό, όπως είπαν και άλλοι, είναι ο τομέας της εκπαίδευση επίσης. Επειδή η οικολογική καινοτομία δεν μπορεί να επιτεθεί παρά μόνο με ικανούς και καταρτισμένους ερευνητές. Αυτά τα λέμε αλλά δεν, έχουμε, δεν έχουμε επεκταθεί λόγω περιορισμένου χώρου. Μόνο στην παράγραφο 5, η παράγραφος 5 μάλλον δεν με ενισχύει βέβαια ιδιαίτερα, μου φαίνεται κάπως παράτολμη, κάπω φιλόδοξη. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις μόνο με την οικολογική καινοτομία. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε εδώ μάλλον μια διατύπωση, θα έλεγα, ίσως πιο μετριοπαθή. Όπως είπα όμως, ο τομέας της εκπαίδευσης, της περαιτέρω κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας, όλα αυτά είναι σημαντικά για την εξασφάλιση και της απασχόλησης. Συνολικά μου φαίνεται σωστό το σχέδιο και ασφαλώς θα το υποστηρίξουμε μόνο ορισμένα θέματα θα προσθέσουμε ακόμα κάποιες πτυχές, σε ορισμένα θέματα δηλαδή. Ο κ. Σέρκας. Εξ ονόματος ε, της συναδέλφου King Gáns που βρίσκεται σε άλλη επιτροπή και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, ε, ζητά συγγνώμη. Θα ήθελε να σχολιάσει το κείμενο του Φιλ Μπενιών, το οποίο δεν μας θέτει κανένα πρόβλημα, αλλά ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία που λείπουν και γι' αυτό θα υποβάλουμε τροπολογίες. Βεβαίως έχει μεγάλη σημασία η εκπαίδευση και η κατάρτιση και πρόθεσμα και όχι μόνο πρόθεσμα. Έχει μεγάλη σημασία για, τους, για τις γυναίκες και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Η λέξη ποιότητα δεν υπάρχει στη γνωμοδότηση και νομίζουμε ότι η καινοτομία και το μέλλον βασίζονται στην ποιότητα, όχι τόσο πολύ στο κόστος, αλλά στην επιστήμη και την ποιότητα. Ε, αυτή αυτή η καιρή καιρή ενώπιον μας ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να συντονιστούμε όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά να υπάρχει συνεργία μεταξύ τεχνολογικών Ινστιτούτων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Και τέλος, αν και ελέγχθη και αλλού, αυτές οι νέες ευκαιρίες και προκλήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται στην αυτή πραγματικότητα των τοπικών αρχών, των επιχειρήσεων και όλων των τομέων, γιατί πρόκειται για μια δύσκολη μετάβαση και δεν θα πρέπει να επαφιέμεθα μόνο στις δυνάμεις της αγοράς, έτσι ώστε να επιβιώσει ο ισχυρότερος. Θα πρέπει δηλαδή να συνοδεύουμε αυτά τα μέτρα, να δούμε ποιοι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση και να τους στηρίξουμε. Να δούμε δηλαδή την πραγματική οικονομική κατάσταση για αυτή την μετάβαση έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν να παρέμβουν. Όχι, η Επιτροπή, ο κύριος Μαρτά. Donc, euh, Η Επιτροπή θα ήθελε να αναφέρει ότι εκτιμά αυτή την έκθεση, η οποία έχει πραγματικά, πραγματιστικά στοιχεία, είναι ε, σαφής και σύντομη και για να μιλήσουμε για την οικοκαινοτομία και το συσχετισμό με την απασχόληση, ε, μία αποτίμηση που έχει αναλάβει ο εκτελεστικός φορέας για την ανταγωνιστικότητα στην ε, Ευρώπη, ένα ε, πρόγραμμα επίδειξης για την οικογενοταμία δείχνει ότι μετά από κάθε πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται δημιουργούνται 8 σταθερές θέσεις εργασίας μετά από 5 χρόνια είναι ένα αριθμητικό στοιχείο το οποίο δεν ισχύει παντού, αλλά υπάρχει αυτή η αιτιώδη συνάφεια. Υπάρχει λοιπόν, ε, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, το ευεργέτημα αφορά όλους και κάτι άλλο που αφορά την καινοτομία θα πρέπει να ε, χρηματοδοτηθεί στο ύψος των ε, φιλοδοξιών που έχουν ε, εκφραστεί. Σας ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν άλλοι που ζητούν το λόγο, δίνω πάλι το λόγο τον, στον Φιλ Μπενιόν για να ολοκληρώσει. Ε, καλωσορίζω όλα τα σχόλια τα οποία λάβαμε και είμαι σίγουρος ότι οι σκιώδεις θα μπορέσουν να διευρύνουν κάπως το πεδίο εφαρμογής και να βελτιώσουν τα στοιχεία μας. Πάντα βεβαίως ε, υπάρχουν περιορισμοί, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε να σταθούμε ε, επί της ουσίας. Από εκπαιδευτικής πλευράς θα ήθελα να πω ότι συνεργάζομαι με τους ε, συναδέλφους οι οποίοι ε, ακριβώς έχουν αυτό το όραμα της εκπαίδευσης ε, πίσω από την οικοκαινοτομία και συνεργάζομαι με έναν συνάδελφο για την εκπαιδευτική πτυχή αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέχρι τις 2 Ιουλίου, θα τις εξετάσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου, ε, μετά στις 18 θα ε, τις εξετάσουμε και θα τις ψηφίσουμε. Και η ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου. Φτάνουμε λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το 18. Πρόκειται για γνωμοδότηση επί της Επιτροπής, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σε σχέση με την εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και έλεγχο των κρατών μελών για την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Οι συντονιστές ζήτησαν να σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχετε λάβει λοιπόν το σχέδιο αυτό που σχετίζεται με τις δεσμεύσεις μας ε, που είναι περιοριστικής υφής τη στιγμή που σε σχέση μάλλον με το αρχικό κείμενο και θα ήθελα να επιμείνουμε επί ορισμένων βασικών αξώνων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, σημασία που προσδίνουμε ως Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση σε σχέση με τις ε, εκτελεστικές αρμοδιότητες στο πολιετές πλαίσιο και επίσης η εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λάβει υπόψη τη σημασία αυτών των θεμάτων από πολιτικής και στρατηγικής πλευράς. Είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε διότι στα πλαίσια της ε, έκθεσης της Utah Steinruth ασχολούμεθα με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις στα πλαίσια της έκθεσής της για την ε, κοινωνική ευρωπαϊκή καινοτομία. Ε, προς υπόμνηση η διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου στα πλαίσια του πολιετούς πλαισίου ορίζει ότι οι στόχοι και οι προτεραιότητες καθώς και οι δημοσιονομικές πρικοδοτήσεις θα πρέπει να εγκριθούν ε, με εκτελεστικές, ε, με, με κατεξουσιοδότηση συγγνώμη, ε, πράξεις και με βάση τις βασικές νομοθετικές αρμοδιότητες. Εξάλλου σας προτείνω να επικρίνουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο, όχι χάρην επίκρισης, αλλά διότι τα δύο αυτά θεσμικά όργανα αποφεύγουν συστηματικά την προσφύγη σε κατεξουσιοδότηση πράξης, υποστηρίζοντας προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό οδηγεί σε ε, ένα ε, νομοθετικό μπλοκάρισμα. Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν λαμβάνουν υπόψη το πνεύμα των άρθρων 290-291 των συνθήκων, όπου προσδίδουμε, προσδίδουμε ξεχωριστό χαρακτήρα στις κατεξουσιοδότηση πράξη σε, σε σχέση με τις εκτελεστικές πράξεις. Και θα ήθελα Θέλω το Κοινοβούλιο να αμφισβητήσει το κύρος των πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν δεν περιορίζεται στα πλαίσια, στις πραγματικές ε, αρμοδιότητες εκτέλεσης όπως ισχύει στην απόφαση Γιούρες και ζήτησαμε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να προσφύγει στο ΔΕΚ σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σε κατεξουσιοδότηση πράξης και θα ήθελα να ότι τώρα εξετάζει το θέμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ίσως αποφανθεί στο τέλος της θητείας στα πλαίσια της ευθυγράμμισης των παλαιών μέτρων επιτροπολογίας και εκείνων που έχουν ε, υποβληθεί σε ρύθμιση με έλεγχο, την λεγόμενη διαδικασία ΠΡΑΚ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με κατεξιοδότηση πράξης. θα θέλαμε να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, της γενικότερης διαπραγμάτευσης και θα θέλαμε η Επιτροπή και το Συμβούλιο να λαμβάνει υπόψη της κατεξιοδότηση πράξεις που δεν λάβαν υπόψη ιδιαίτερα στα πλαίσια του φακέλου της υπόθεσης Γιούρες. Σας ε, παρουσίασα το περιεχόμενο αυτής της γνωμοδότησης και είμαι στη διάθεσή σας για να συμπληρώσετε αν θέλετε, αν το επιθυμείτε. Ποιος ε, ζητά το λόγο παρακαλώ. Βλέπω ότι πολύ σας ε, παθιάζει αυτό το θέμα. Εντάξει, ε, το καταλαβαίνω, αλλά είναι θέμα εξουσιών της Επιτροπής μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Γιατί το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια κινητοποιείται στα πλαίσια της Επιτροπολογίας, ώστε να μην παρακάμπτεται στην απόφαση. εξαιτία των κατεξοδότηση πράξεων που έχει η Κομισιόν. Καλά, αν δεν έχετε σχόλια, τότε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών, που θα είναι πολλές, σίγουρα 26 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Θα τις εξετάσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Εδώ, 25 και 26 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα αποφανθεί επί της έκθεσης του κ. Σιάγερ 9 ή 10 Οκτωβρίου. Πάει και αυτό το σημείο. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 19. Εδώ έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής μας για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισαγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών και συναφή μέτρα. Πρόκειται εδώ για την ποσόστοση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, έτσι. Η Επιτροπή Γυναικών είναι επίσης αρμόδια επί της ουσίας από κοινού με την Νομική Επιτροπή. δικιά μας εισηγήτρια είναι η κυρία Μαρέγια Κορνέλισεν και της δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει τις 167 τροπολογίες 42 δικές της μάλιστα που υποβλήθηκαν επί του σχεδίου αυτού γνωμοδότησης. Έχετε το λόγο κυρία Κορνέλισον. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους σκιώδεις και όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Υπάρχουν ε, διαφορές απόψεων, δεν μας εκπλήσει αυτό. Σε πολλά όμως υπάρχει συμφωνία, υπάρχουν πολλές καλές ιδέες. Πολλοί από εμά εδώ στο Κοινοβούλιο όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και έτσι έχουμε και πιο πολλές πιθανότητες να περάσει ο δικός μας λόγος στο Συμβούλιο. Κοιτάξτε, έφτιαξε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε όλοι. Αυτό εδώ το χρωματιστό σχεδιάγραμμα. Πριν από μερικούς μήνες ή εβδομάδες ήμουν σε ένα αεροπλάνο και ξαφνικά σκέφτηκα, μα πρέπει να καταλάβω καλύτερα Πώς γίνεται αυτό ακριβώς το θέμα στα διάφορα κράτη-μέλη και σε επιχειρήσεις. Και γι' αυτό όπως ήμουν στο αεροπλάνο σκέτσαρα κάτι, έφτιαξα κάτι και το έδωσα και στους συνεργάτες μου που το προχώρησαν και το βελτίωσαν. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ και με τα σχόλια που είχε κάνει ο κύριος Φιλ Πενιον την τελευταία φορά που το συζητήσαμε. Αριστερά πάνω βλέπετε το κράτος μέλος που πρέπει να αξιολογήσει τα μέτρα που έχει, αν έχει. Αν έχει, μπορεί να ζητήσει άρση για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε πολιτική που έχει. Εφόσον τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι θα καταλήξουν στο σωστό αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Η πρόοδος βέβαια το 2017 θα εκτιμηθεί. Εάν η πρόοδος είναι επαρκής, οδηγεί σε επιτυχία. Αν δεν είναι επαρκής η πρόοδος ή το κράτος μέλος ζητάει να μην υπάρξει άρση, δεν έχει καθόλου μέτρα, τότε θα πρέπει να εισάγει νομοθεσία. Αν δεν το κάνει, πρόκειται για παραβίαση, επιβάλλονται κυρώσεις Αυτά είναι συνηθισμένα για όλες τις ευρωπαϊκές οδηγήσεις και αυτό. Οι επιχειρήσεις τώρα πρέπει να αξιολογήσουν αν έχουν 40% και από τα δύο φύλλη. Αν έχουν, το καλύτερο. Αν δεν έχουν, τότε πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους. Αν ναι, τότε είτε έχουν καλά αποτελέσματα ή όχι. Αν έχουν καλά αποτελέσματα, τόσο το καλύτερο. Αν όχι, πρέπει να εξηγήσουν τι συνέβη και να πάρουν μέτρα. Στην οδηγία προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι. Για μια επιχείρηση η οποία πάει καλά, έχει αποτελέσματα, τότε η υποχρέωση αναφοράς της επιχείρησης αυτής θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ελαφρά. Αν όμως τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, τότε βέβαια επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η αναφορά αυτή της επιχείρησης. Αν το αποτέλεσμα είπαμε είναι εντάξει, έχει καλώς, αν δεν είναι πρέπει να πει γιατί και να πάρει μέτρα. Αυτός είναι βέβαια ένας φαύλος κύκλος κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κάθε φορά που δεν έχει επιτυχία συνεχίζεται το ίδιο. Αν τώρα μία επιχείρηση αρνηθεί να προσαρμόσει τις διαδικασίες της ή αρνηθεί να εξηγήσει και να πάρει μέτρα, τότε έχει κυρώσεις. Κυρώσεις δεν είναι αν δεν έχει πετύχει το 40%, είναι αν δεν κάνει τίποτα. Ελπίζω με το σχεδιάγραμμα αυτό να καταλαβαίνετε καλύτερα ότι οι χώρες μέλη τιμωρούνται εφόσον δεν κάνουν τίποτα και επιχειρήσεις επίσης έχουν κυρώσεις μόνο εάν δεν κάνουν τίποτα. Αν προχωράνε έχουν αποτελέσματα είτε τα κράτη-μέλη με την πολιτική τους είτε επιχειρήσεις, τέλεια. Ελπίζω το σχεδιάγραμμα αυτό να σας βοηθήσει. Τώρα θέλω να κάνω παρατηρήσεις για μερικέ τροπολογίες. Την επόμενη εβδομάδα στη συνάντηση σχεδόν, θα συζητήσουμε το εύρο εφαρμογή κατά πόσο πρέπει να επεκταθεί στι μικρομεσαίε που είναι εισαγμένε ή σε όλες τις εισαγμένε ή σε όλες τις μη εισαγμένε επίσης ή αν αντίθετα πρέπει να περιορίσουμε το θέμα αυτό να μην συμπεριλαμβάνονται μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις από αυτού που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό που, προστα... που προστέθηκε εδώ. Διαφάνεια, οικογενειακή ζωή. Τη διαφάνεια ο κύριος Λούτβικ. Την έβαλε ο ορισμός πώς γίνονται οι ορισμοί και τη συμμετοχή των μετόχων και πώς να χειριστούμε τις κυρώσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο τι κυρώσεις θα επιβάλλουμε ή είναι τα κρατη που τις αποφασίζουν. Αυτά προς το παρόν και περιμένω να ακούσω τι έχουν να πούν οι άλλοι σκιώδεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σάγια. Αντικαθιστάτε νομίζω την Ερυμπάουερ και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, η συνάδελφός μου δεν μπόρεσε να προσέλθει. Ζητεί συγγνώμη λοιπόν για την απουσία της και θα παρουσιάσω τις δικές της απόψεις, οι δικές μου αποκλίνουν λίγο, αλλά αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Πρώτα λοιπόν θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της προτάσεως οδηγίας νομίζει ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε έστω και αν υπάρχει νομοθεσία η οποία ε, στοχεύει στην κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων, εξακολουθούν να υπάρχουν οι διαφορές και διακρίσεις αυτές. Τώρα η Κομισιόν προτείνει την ελόγω ε, νομοθεσία για να βελτιώσει την κατάσταση στον επιχειρηματικό τομέα. Η συνάδελφός μου Χαίρεται για το γεγονός ότι η Κομισιόν προσπαθεί να τηρήσει την αναλογικότητα στην πρόταση και θεωρεί ότι πρέπει να πράξουμε πάντο δυνατό για να συμβάλλουμε στην γέννηση αυτής της νέας οδηγίας και να μην ε, υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες να την φρενάρουν όπως έχουμε, έχουμε δει σε άλλους φακέλους, σε άλλα θέματα. Θεωρεί ότι η Κομισιόν έκανε καλά, παρέμεινε μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας και θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Γνωρίζει ότι το Συμβούλιο δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι απαιτείται η νομοθεσία αυτή. Έτσι λοιπόν, εποφελία των ψηφοφόρων μας, ας φτιάξουμε οδηγία η οποία να καθορίζει την θέση των γυναικών μέσα, στα επιχειρηματικά, μέσα στις επιχειρήσεις. Η συνάδελφός μου θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή της πρότασης της Κομισιόν ώστε στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, να περιληφθούν μόνο οι εισηγμένε εταιρείε και οι εισηγμένε δημόσιε επιχειρήσει. Ωστόσο, ο συνάδελφό μου δεν είναι υπέρ τη συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αν και ορισμένοι συνάδελφοί μου εξέφρασαν τέτοιε προθέσει. Επίση, υποστηρίζει την θέση τη Κομισιόν στην προσπάθεια επίτευξη ενό 40% γυναικών μέσα στα πλαίσια των Συμβουλίων και εν πάση περιπτώσει ένα τρίτο όλων των θέσεων διευθυντών ανεξαρτήτως του εάν είναι εκτελεστική ή μη εκτελεστική η ε, υπάλληλη αυτή. Λέει όμως ότι πρέπει να περιληφθούν όλοι και σε όλα τα επίπεδα. Εν τέλει θεωρεί ότι θα πρέπει πρωτίστως να αναμένουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας σχετικά με τη νομική βάση της οδηγίας. Ε, Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ήδη συζητήσαμε μετά την κατάθεση του σχεδίου γνωμοδοτήσεως και θα επαναλάβω τα ίδια. Έχω να πω τα εξής. συμφωνώ σε πολλά και με τα σχόλια της κυρίας Μπάουερ. Να είμαστε φιλόδοξες, αλλά ταυτόχρονα να ε, ε, φροντίσουμε να υποβάλουμε ένα τελικό κείμενο το οποίο να μπορεί να γίνει και αποδεχτό και από ανθρώπους που έχουν ίσως κάπως διαφορετικές απόψεις. Προσωπικά δεν συμφωνώ να μπουν μέσα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω βάλει αρκετές τροπολογίες που λέω ωστόσο μιλώ για ενθάρρυνση και χορήγηση κινήτρων για εκτελεστικούς και μη ε, διευθυντές ή ε, διευθύνοντες συμβούλους στην περίπτωση αυτή. Ε, νομίζω ότι στα πλαίσια της γνωμοδότησης, τουλάχιστον στις αιτιολογικές σκέψεις, πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα μιας ισορροπίας των φύλων, των στελεχών που λαμβάνουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα μιας επιχειρήσεως. Γιατί καμιά φορά οι γυναίκες επικρίνονται για το γεγονός ότι εάν έχουμε έναν αριθμό γυναικών μέσα σε κάποια συμβούλια. Αυτό αρκεί για την εξασφάλιση τη ισότητα των φύλων. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, δεν αρκεί. Πρέπει να δούμε τι γίνεται σε όλα τα επίπεδα τη επιχείρηση, ώστε να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν όργανα λήψη αποφάσεων με ισορροπία φίλων. Επίση, αναφέρθηκα και στα θεσμικά όργανα τη Ένωση τη τροπολογία μου. Δεν ξέρω αν τα έχει σκεφτεί κανεί αυτά. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουν την πρόταση αυτή, ασφαλώς και θα πρέπει πρωτίστως να εξετάσουμε τα του οίκου μας και να μην προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να εφαρμόσουμε τα όσα περιλαμβάνει η οδηγία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει να περιληφθεί έστω και στις αιτιολογικές σκέψεις. Όπως είπα, έχω καταθέσει ορισμένες τροπολογίες που ενθαρρύνουν και προσφέρουν κίνητρα και σε επιχειρήσεις και στις χώρες μέλη, έτσι ώστε να θεσπιστούν από τις χώρες μέλη πιο ευνοϊκές διατάξεις από αυτές που ανταποκρίνονται αυστηρά στο περιεχόμενο της οδηγίας. Μιλώ και για διαφάνεια κλπ. Ελπίζω θα έχουμε, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να διαβουλευτούμε περισσότερο και να καταθέσουμε κοινά αποδεκτές τροπολογίες. Ευχαριστώ. κυρία Ρέγκνερ. Ευχαριστώ κυρία Παρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά την εισηγήτρια και ιδίω το έγχρωμο αυτό σχέδιο. Πάντως ομολογώ ότι είμαι, μου αρέσει μεν χρωματικά, αλλά ε, τελώ σε κάποια σύγχυση. Ίσως να κάνουμε μια προσπάθεια να το απλοποιήσουμε. Πάντως η κατεύθυνση που λαμβάνεται είναι σωστή ένα σύντομο σχόλιο. Αύριο το πρωί στην νομική υπηρεσία και στην υπηρεσία και στην νομική επιτροπή και στην Επιτροπική Διωμάτων Γυναικών έχουμε ενδιαφέρουσα ακρόαση με εθνικούς και εθνικές βουλευτές που έχει ενδιαφέρον να περιγράφουμε δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο στις συζητήσεις αυτές και του εθνικούς βουλευτές διότι η συζήτηση αυτή διεξάγεται με αρκετό πάθος και στις χώρες μέλη και είναι αρκετά ανάγλυφη η εικόνα της καταστάσεως. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, διότι υπάρχουν πολλές και ποικίλε απόψεις. Πάντως, το σεμινάριο που είπα ήταν ενδιαφέρον. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της σκιώδησης εισηγήτριας Βίνκελ που είναι Λιθουανή και είναι ενθουσιώδης υπέρ του θέματος Επίσης θέλει να το περιλάβει στην ημερήσια διάταξή της και η Λιθουανική Προεδρία. Τα πιο σημαντικά της σχόλια εν προκειμένου είναι τα εξής τρία. Πρώτα, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σχετικά με το αν θα πρέπει να περιληφθούν ή όχι. Προτείνει να επεκταθεί η, το επαιδείο εφαρμογή της οδηγίας και σε μη εισηγμένε δημόσιες επιχειρήσεις, διότι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να περιληφθούν στα συμβούλια των ε, μη εισηγμένων δημόσιων επιχειρήσεων γυναίκες. Ορισμένες χώρες μέλη ήδη εγκύπτουν στο θέμα, ιδίω λοιπόν για τις δημόσιες επιχειρήσεις, όπου πάνε να δώσουν το καλό παράδειγμα. Αυτό λοιπόν θα ήθελε να περιληφθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την επέκταση ώστε να καλυφθούν και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να λεχθεί απλά ότι θα πρέπει να είναι σε πρωτοπόρα θέση και να περιληφθούν επομένως στην οδηγία, ώστε <clears throat> οι συγμένες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους στόχους της οδηγίας λόγω της οικονομικής τους βαρύτητας και της βαρύτητάς τους όσον αφορά την απασχόληση και η κυρία Δικεβιτσιούτε θέλει να αναφερθεί και στην καταληκτική ημερομηνία της οδηγίας που βρίσκει ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξη. Δεν νομίζει ότι θα επιτύχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Προτείνει λοιπόν κατάργηση της καταληκτικής ημερομηνίας διότι θεωρεί και όλος ότι το θέμα αυτό δεν επιδέχεται τέτοιους περιορισμούς. Εν τέλει το ζήτημα των κυρώσεων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εφαρμογή κανόνων αν δεν προβλέπονται κυρώσει, Αυτό είναι σίγουρο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι αποτελεσματικό, αναλογικός και προοδευτικό. ο κανόνα. Οι κυρώσει δηλαδή. Οι κυρώσει δεν θα πρέπει να λένε may αλλά shall. Μετά από ε, πρώτες ε, προειδοποιήσεις θα πρέπει να ακολουθούν κυρώσει που θα επιβάλλονται από δικαστικό όργανο. Αυτά είναι ολίγης η σκιώδη συγκεκριά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τάσεται υπέρ της οδηγίας, η οποία και αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο δεσμευτική. Εγώ ως εισηγήτρια στην Νομική Επιτροπή ε, έχω κάποια κατανόηση για τα σχόλια που θα ήθελε η ίδια να περιληφθούν. ευχαριστώ πολύ. Φιλίπ Μπενιό. Και παραμένουμε εκεί. Να απαντήσω στην κυρία Κορνέλησαν επειδή απευθύνθηκε σε μένα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πιο εμπεριστατωμένο πλαίσιο αυτό που βλέπετε εδώ. Ε, βεβαίως δεν έχουμε διαρθωτικά προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, αυτές τις τυχές διακρίσεις και αυτό είναι πολύ καλύτερο. Εγώ δεν νομίζω ότι οι ε, ποσοστός όπως ορίζονται ε, είναι σωστές. Ως προς την γραφική παράσταση θα ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν πάντα νομοθεσία. Ίσως χρειαζόμαστε ε, μη, ίσως πρόκειται για μη νομοθετικές ελλείψεις και δεν χρειάζεται ε, νομοθεσία ή νομοθέτηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δεν ε, νομοθετεί στο κράτος τότε υπάρχει παραβίαση. Νομίζω ότι η νομοθεσία ε, είναι καλή, κάλλιστη, αλλά δεν είναι και η μοναδική λύση. Θα πρέπει να προωθήσουμε και την εκπαίδευση και την κατάρτιση προς τις σωστές κατευθύνσεις και τους σωστούς ανθρώπους. Άρα το θέμα δεν είναι καθαρά νομοθετικό. Ως προς τις εταιρείε κάθε αυτές μπορεί να, κάνουν, να τα κάνουν όλα και να μην φτάσουν στο 40%. Αυτό μπορεί να είναι τομεακό καθαρά. Δηλαδή να αφορά τα καλλιντικά ή ορισμένους τομείς όπου δεν υπάρχουν αρκετές ε, προσλήψεις. Άρα μπορείτε στο δινικές να βρίσκεστε, να βρίσκεστε σε αυτή τη θέση. Αν το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να δεχτούμε, ακόμα και αν γίνουν ε, σωστά όλα, ίσως η έκβαση να μην είναι αυτή που επιθυμείτε πάντα. Υπάρχει κάποιος από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε το λόγο όχι να μας πει ότι είναι εξαιρετικό το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Μιχαήλ Γκόντε από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης δεν έχουμε ιδιαίτερα σχόλια για τη συζήτηση. Η κυρία Κορνέλισεν έχει το λόγο. για τον κύριο Μπάνιον. Πολύ σωστό αυτό που είπε για την νομοθεσία θα το αλλάξω στον πίνακα γιατί δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ένα νομοθέτημα ή άλλα μέτρα. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι ακόμα κι αν μία επιχείρηση έχει, τα έχει, έχει όλα τα στοιχεία σωστά, ίσως είναι κάπως ε, στριμωγμένη ή παραμείνει στριμωγμένη στο δινεκές. Είπα και σε κάποιον άλλον, το είπα και αλλού αυτό και μίλησα για μία επιχείρηση όπου ας πούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο κάποιος που φέρει ένα συγκεκριμένο όνομα μπορεί να βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν γυναίκες και πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ως προς τα άλλα σχόλια, η κυρία Εσάια με βρίσκει σύμφωνη ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την οδηγία για να την καταστήσουμε πιο σαφή ε, για τα κρατη δηλαδή να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά να μπορέσουμε να περάσουμε και τη θέση μας ε, στο Συμβούλιο. Βεβαίως είναι μια ε, γνωμοδότηση προς τη Γιούρη και τη ΦΑΜ. Έχουμε περιθώρια δηλαδή να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι. Συμφωνώ με την Μάριον Χάρκιν ότι θα θέλαμε να εντάξουμε πολλά στοιχεία, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό αφορά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μπορούμε να, το, να αναφερθούμε στην αιτιολογική σκέψη έτσι ώστε να είμαστε πιο ε, αξιόπιστοι προς τον ε, εξωκόσμο, να μην υπάρχουν ε, διακρίσεις ως προς το φύλλο. Το θέμα του πεδίου εφαρμογής θα το συζητήσουμε με τους κοιόδης. Ας αφήσουμε τη νομική βάση στη Γιούρη που είναι η Επιτροπή επί της ουσίας και μπορεί να το συζητήσει. Δεν θα ήθελα να μας απασχολεί στην Επιτροπή Απασχόλησης. Για τα υπόλοιπα θα ε, αντιδράσω αργότερα στην ε, συνάντηση σκιωδών, αλλά νομίζω ότι θα είναι συνενετική αυτή η γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε θα εξετάσουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού 8 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε στις 9 του μηνός οι Επιτροπές Φάμα και ε, Νομικών Υποθέσεων στις 16 και 18 Σεπτεμβρίου θα γνωμοδοτήσουν. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. περνάμε στο σημείο 20. Σχέδιο γνωμοδότηση του συναδέλφου Ταμάς Deutsch Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Πρόκειται για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων διαδικτύου οργανισμών του δημόσιου τομέα. Αλλά θα αντικαταστήσει ο κύριος Κοζά τον κύριο Deutsch. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, ο συνάδελφος, ο κύριος Ντόιτσε, λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ, γιατί συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε μια άλλη συνεδρία, σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω τα πιο βασικά στοιχεία της γνωμοδότησής του. Θα αρχίσω από δύο στοιχεία που θέλει να υπογραμμίσει και ο κύριος Ντόιτς. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τα ίδια δικαιώματα για να διασφαλίσουμε μια κοινωνία όπου να συμμετέχουν όλοι, να μην αποκλείεται κανείς. Δεύτερο βασικό στοιχείο για τον κύριο Ντόιτς είναι ότι η προσβασιμότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις μεταξύ τους να προσπαθήσουν να συγκλίνουν. Μιλάμε λοιπόν για την προσβασιμότητα των ιστότοπων, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι και τα άτομα με αναπηρίες και τα πιο ευάλωτα άτομα της κοινωνίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια αγορά που έχει και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Η προσβασιμότητα λοιπόν των ιστοτόπων αντιστοιχεί σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το μέρος της στην αγορά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία να είναι σαφής και να μην επιδέχεται παρερμηνίες. Ο εισηγητής είναι βέβαιος ότι εφόσον η ρύθμιση είναι καλή, τότε όλοι οι χρήστες θα δουλέψουν προκειμένου να επιτευχθεί η προσβασιμότητα αυτή για όλους και θα υπάρχουν και θετικές συνέπειες επί της καινοτομίας. Ο κύριος Ντόιτς έχει παρουσιάσει πολλές τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την προστασία προσωπικών δεδομένων για την ασφαλή μεταβίβαση των δεδομένων και προκειμένου να διευκρινίσει κάποιες έννοιες. Είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικό πριν από οτιδήποτε άλλο να άρουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στην ιστοπροσβασιμότητα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να καταρτήσουμε ειδικού ώστε να καλύψουν ό,τι αδυναμίες και κενά υπάρχουν. Θέλω να επιστήσω επίσης την προσοχή σας στις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για την προσβασιμότητα αυτή, δηλαδή τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις που δεν θα πρέπει να βαρύνουμε με περισσότερη γραφειοκρατία. Η κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ και εγώ τον εισηγητή. Κοίταξα τις τροπολογίες και νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τις περισσότερες από αυτές. Η μόνη που με βρίσκει πολύ σκεπτική είναι η τροπολογία αριθμό 11. Και αυτό γιατί λέει ότι οι ιστότοποι ε, πρέπει να είναι προσβάσιμοι ε, ιδίως για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς συμπεριλαμβάνουν των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων. Δεν ξέρω αν όντω ε, πρόκειται για ομάδα που έχει λειτουργικούς περιορισμούς ή αναπηρίες αλλά ας πούμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό. Πάντως, οι δημόσιοι οργανισμοί που αναφέρονται στο παράρτημα είναι τέτοιοι που πρέπει να τους ξαναδούμε. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλους. Δεν ξέρω τι λέει ο εισηγητής. Στο σημείο 10 αναφέρεται η ανώτατη εκπαίδευση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε για όλη την εκπαίδευση, όχι μόνο για την ανώτατη. Και στο σημείο 1 αναφέρονται οι φόροι εισοδήματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και φόροι ιδιοκτησίας και άλλοι. Η προσβασιμότητα πρέπει να υπάρχει για όλους τους φόρους, όχι μόνο για τους φόρους εισοδήματος. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν. που σημαίνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι τέτοιες που να μην εμποδίζουν την προσβασιμότητα. Άρθρο 9. Η ερώτησή μου είναι σαν και αυτή που ρώτησα και πριν όταν συζητούσαμε την ισότητα των δύο φύλων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αν εδώ θέλουμε να έχουμε ιστότοπους των δημοσίων οργανισμών που να είναι προσβάσιμοι, Ας δούμε πρώτα απ' όλα τις ιστοσελίδες, τους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως και εκεί θα πρέπει να αλλάξει κάτι. Αν μη τι άλλο, ας το συζητήσουμε. Είτε είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, είτε όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Συμφωνώ με τον εισηγητή πάντως για το ότι έχει μεγάλη σημασία η πρόσβαση, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπηρίες. Η προστασία των δεδομένων και η συνέργεια μεταξύ διάφορων εμβληματικών πρωτοβουλειών, άρση των εμποδίων, συμφωνώ με όλα αυτά. Και προσβλέπω και εγώ σε καλή συνεργασία μεταξύ μας για να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Αλεχάνδρου Θέρκας. Ευχαριστώ. Η σκιώδης η συγγήτρια είναι η κυρία Κίνκα Γκόνς και ετοιμάζει τροπολογίες για να συμπεριλάβει στην έκθεση αυτή, να προτείνει. Δεν βλέπουμε προβλήματα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο μακριά. Για να υπογραμμίσουμε, για παράδειγμα, τη σημασία που έχει η έκθεση αυτή και για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Δεν αποτελεί μόνο ένα εργαλείο, ένα μέσο αυτού, αλλά μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι διάφοροι άνθρωποι στις κοινωνίες μας, όπως αυτοί που έχουν αναπηρία οι ηλικιωμένοι, οι όσοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ορεινές περιοχές, δύσκολα προσβάσιμες. Πολλές φορές οι ιστότοποι δεν είναι καλά φτιαγμένοι για όλους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να συμπεριληφθούν όλοι στην προσβασιμότητα αυτή. Το εύρος εφαρμογής ίσως πρέπει να διευρεθεί λοιπόν και σε αυτές τις κατηγορίες και να μην υπάρχει περιορισμός. Εδώ αναφέρονται διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί δημόσιας δίκησης. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι δημόσιες δικήσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά από τους πολίτες. Αν υπάρχει μια νομοθετική πρόταση, είναι ήδη κάτι, αλλά συχνά λείπει εφαρμογή, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές νομοθετικές ε, ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν τίθενται σε εφαρμογή. Πώς λοιπόν θα διασφαλιστούμε ότι και τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Τέλος, στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5 θα έπρεπε να προσθεθεί κάποιος ορισμός για το χρονοδιάγραμμα Κάτι που να είναι ρεαλιστικό όμως, για να ξέρουμε πότε όλα αυτά θα μπορούμε να τα δούμε στην πράξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιος εσείς. Ναι, έχουμε κάποια σχόλια. Πρώτον για την τροπολογία αριθμός 10 όσον αφορά την συμμετοχή των εταίρων στην Συμβουλευτική Επιτροπή. Εκείνη θα αποφασίσει. Το πρόβλημα είναι ότι οι εταίροι δεν μπορούν να συμμετέχουν. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την επιτροπολογία. Μπορεί να υπάρξει διαβούλευση από την Επιτροπή μαζί τους και το φροντίζουμε, αλλά οι εταίροι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες επιτροπές που είναι για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφερόμενοι, μόνο μια σχέση συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορούν να έχουν μαζί μας. Μπορούν να συμμετέχουν στους μηχανισμούς που θα αποφασιστούν για τον έλεγχο της εφαρμογής. Και αυτό αποφασίζεται από τις εφαρμοστικές διατάξεις, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές. Τροπολογία 15 τώρα, για την ενημέρωση του κοινού και τον κατάλογο που υπάρχει στα παράρτημα. Αυτό σημαίνει όλες, όλοι οι ιστότοποι, όλες τις δημόσιες δίκησης. Οπότε συμφωνούμε και με την πρόταση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Όσον αφορά τώρα την υποχρέωση προσβασιμότητας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέτε, υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί δεν εμπίπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί προκειμένου να υπάρχει προσβασιμότητα του κόσμου στις, στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή δεν μπορεί να συμπεριλάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα κάνει να αποτελέσει παράδειγμα και να φροντίσει να είναι η πρώτη που έχει προσβάσιμους όλους τους δικούς της ιστότοπους στον κόσμο. Παρακαλώ. Τώρα, ο συγκητής. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για τις παρατηρήσεις σας. Εννοείται ότι θα μεταφέρω όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας στον κύριο Ντόιτς, που είναι υπεύθυνο. Μία παρατήρηση έχω να κάνω εγώ. Εδώ δεν πρόκειται για γνωμοδότηση περί κατά. Είναι ένα θέμα κέριο. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της υπέρ των ατόμων με αναπηρίες και αυτό για την περίοδο από το 2015 και ξεκίνησε διαβούλευση μέσω του διαδικτύου. για τη στρατηγική ακριβώς αυτή για τα άτομα με αναπηρίες. Ελάχιστα πράγματα αναφέρθηκαν στο διαδίκτυο. Και γιατί, γιατί ακριβώς τα άτομα με αναπηρίες δεν είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο για να μεταφέρουν τις απόψεις τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Πρόεδρο ευχαριστούμε τον εισηγητή. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 2 Ιουλίου. Θα τι εξετάσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου και θα εξεταστούν στις 27 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 26. ΙΜΚΟ θα αποφανθεί 27 και 28 Νοεμβρίου. Τώρα. Η κυρία Σιπέλη είναι η επόμενη εισηγήτρια για το επόμενο θέμα. Η κυρία Κίνγκα Κοντσέτσι κι αλλιώ είναι στη Λίμπε και ψηφίζει, οπότε προτείνω να αντιστρέψουμε τα σημεία 21 και 22. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Σκριντεύσκα, οποία θα μας παρουσιάσει τις 331 τροπολογίες, οι οποίες υποβλήθηκαν στην έκθεση πρωτοβουλίας της για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Πιθανές λύσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μια ίδια πρωτοβουλία, όπως είπατε κι εσείς. Όντω 337 πρωτοβουλί... ε, τροπολογίες υποβλήθηκαν. Σας ευχαριστώ όλους και κυρίως τους ευρωβουλευτές εκείνους που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή. Για μένα το ότι οι τροπολογίες είναι τόσο πολυάριθμες αντικατοπτρίζει το γεγονό ότι Όλοι ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο λύση. Οι περισσότερες τροπολογίες που υποβλήθηκαν πάντως θα τις δεχτώ. Είναι τέτοιε που θα τις δεχτώ. Εδώ δεν θα αναφερθώ σε κάθε μία χωριστά γιατί θα είμαστε ακόμα εδώ την επόμενη εβδομάδα. Αυτό όμω που θέλω να κάνω είναι να αναφερθώ στις τροπολογίες εκείνες για τις οποίες έχω κάποιες αμφιβολίες. Και θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Με την έκθεση αυτή θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση των νέων που δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημερινή οικονομική κρίση. Εννοείται ότι η οικονομική κρίση είναι το κερασάκι στην τούρτα και είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Αλλά είναι και διαρθρωτικό το πρόβλημα. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, για να ζητήσουμε από τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν περισσότερο και με την κατάρτιση και έτσι να πάψει αυτό το πρόβλημα που είναι ότι η κατάρτιση, η εκπαίδευση των νέων δεν τους προσφέρει τα κατάλληλα προσφόντα για να μπορέσουν να απασχοληθούν στις επιχειρήσεις. Δεν έχουν αρκετή εμπειρία. Ας αποκτήσουν εμπειρία και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Να συμμετέχουν επιχειρήσεις σε αυτό. Οι τροπολογίες που αναφέρονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για παράδειγμα, και που λένε ότι θέλουν να διασφαλιστεί αξιοπρεπής εργασία κτλ. Τέτοιου είδους τροπολογίες που αναφέρονται σε που μπορεί να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τίποτα. Ναι, η κοινή γνώμη φυσικά και περιμένει από μας κάτι να κάνουμε δηλώσεις. Αλλά δυστυχώς, δυστυχώς, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι. Οι αρνητικές συνέπειες της μετανάστευσης των νέων είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οι χώρες οι οποίες έχουν περισσότερη δουλειά είναι εκείνες που υποδέχονται και περισσότερους νέους. Οι νέοι, όμως αυτοί ποιοι είναι, αυτοί που είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Πρέπει να ξέρουμε ότι η μετανάστευση αυτή μπορεί να είναι καλή λύση για αυτούς που θέλουν πραγματικά να φύγουν από τη χώρα τους, που στη χώρα πρόλευση τους δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Δεν μπορούμε επίσης να υποσχεθούμε στους νέους ότι μετά από μια άσκηση θα έχουν και μια μόνιμη θέση εργασίας. Δεν υπάρχουν πια τέτοιες πρακτικές, ούτε υπάρχει καμία νομική διάταξη που μπορεί να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα μπορούν να το έχουν αυτό. Δεν μπορεί κανένας επιχειρηματίας να τους εγγυηθεί μια θέση απασχόλησης μετά από μια άσκηση. Αυτό που μπορεί να τους διασφαλίσει όμως είναι τη γνώση που τους προσφέρει, την εμπειρία που τους προσφέρει και η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει στο να βρούνε και μια πιο μόνιμη θέση. Αλλά η πρακτική αυτή θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Θα πρέπει πραγματικά οι νέοι να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της εργασίας και έτσι να γίνουν πιο ελκυστικοί για την αγορά εργασίας φεύγοντας από μια πρακτική σε μια επιχείρηση, ναι, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και την εμπειρία που τους χρειάζεται για να μπορέσουν να βρουν ε, δουλειά. Να έχουν αρκετές εμπειρίες και αρκετή γνώση για να μπορέσουν να σταθούν σε μια νέα θέση απασχόλησης. Τώρα για την διευκόλυνση στην ε, κινητικότητα, για τα δικαιώματα που πρέπει επίσης να μεταφέρονται. Στόχο μας δεν πρέπει να είναι η διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε για την εκπαίδευση σε όλε τις χώρες μέλη και λέμε ότι πρέπει να είναι δωρεάν. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές όμως στις χώρες μέλη. Πρέπει να αποφύγουμε την εξοικονόμηση πόρων από την εκπαίδευση και αν πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί να μην είναι πολλοί. Έτσι κάπως σύντομα σκιαγράφησα τα πιο σημαντικά σημεία. Πραγματικά ήταν μεγάλη χάρα για μένα που μπόρεσα να συνεργαστώ με τις κέντρες συζυγήτρες στην έκθεση αυτή. Είμαστε στη πρώτη τελευταία συνάντηση. Προσπαθούμε να πετύχουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα ξαναβρεθούμε την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε έτσι να συντάξουμε και συμβαστικές τροπολογίες. Το κείμενο δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να είναι σαφές, ευθύ. Ευχαριστώ όλους τις ομάδες, τους ευρωβουλευτές και είμαι πεπισμένη ότι θα πετύχουμε συμφωνία ακόμα και αν προερχόμαστε από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε για την μέχρι τώρα συνεργασία. Όπως εξηγήσατε και εσείς, έχουμε ήδη εξαγάγει μια συνεδρίαση των σκιωδών που πήγε καλά. Αν και βεβαίως δεν διεξήλθαμε όλα ακόμα τα επίμαχα θέματα. Πριν προχωρήσω στις επιμέρους τροπολογίες, και εξηγήσω πού αντιμετωπίζουμε προβλήματα και πού τα πάμε καλύτερα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια ψηφίσαμε ψήφισμα και ότι σε αυτό το ψήφισμα σημειώνουμε καθαρά ότι η απασχόληση των νέων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί να προωθηθεί παρά μόνο μέσα σε μακροοικονομικό πλαίσιο. Άρα εδώ πρέπει να βάλουμε σωστά τι μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Βεβαίως να ληφθούν υπόψη και τα διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως όμως η οικονομική κρίση. Βεβαίω αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά, αλλά εγώ προέρχομαι από μια χώρα, την Αυστρία εννοεί, όπου με το ξέσπασμα της κρίσης το 2008, τα κονδύλια για την ενεργό πολιτική απασχόληση των νέων διπλασιάστηκαν εν μια νυχτή και έχουμε τώρα αποτελέσματα. Δηλαδή το να δώσει, το να ρίξει κανείς χρήματα στην εξασφάλιση απασχόληση των νέων είναι θετικό, είναι διασφάλιση για το μέλλον. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το εθνικό επίπεδο, αλλά και ιδίω για το ευρωπαϊκό. Τώρα για τις τροπολογίες. Τις χωρίζω τώρα ανάμεσα σε αυτές που είναι καταπληκτικές, άλλες που είναι λιγότερο καλές και άλλες που θα χρειαστεί να βρούμε κάποιες συμφωνίες. Όλες οι τροπολογίες για την συμπερίληψη των διαφόρων φορέων, των παικτών και των επιχειρηματιών επομένω. Επίσης, κατάρτιση, εκπαίδευση, οργανώσεις νέων, η δραστηριοποίηση των αρχών σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό κτλ επίσης ιδίως των κοινωνικών εταίρων. Αυτές οι διατάξεις είναι πολύ σημαντικές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τις συγχωνεύσουμε όλες ώστε να καταδείξουμε την ευθύνη που έχουν όλοι οι φορείς. Δεν είναι δυνατόν να λέμε το κράτος έχει ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη. Θα λειτουργήσουν τα πράγματα μόνο με απόλυτη συνεργασία και βέβαια με συνειδητοποίηση της ευθύνης του καθενός φορέα. Όπως είπα επίσης αρχικά, χρειαζόμαστε περισσότερο περισσότερα χρήματα. Τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολογίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας μου φαίνονται εύλογοι, εύλογο ποσόν. Τώρα η σημασία του διτού συστήματος εκπαίδευσης. Πρέπει να τονιστεί αυτό. Γιατί αυτά βάζουν τις βάσεις για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν είναι άμεσα πυροσβεστικά μέτρα, είναι όμως σημαντικές οι τροπολογίες αυτές για να περιληφθούν εδώ και βέλτιστες πρακτικές. Είναι απαραίτητο αυτό για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι μας. Τέλος, η κοινωνική εταίροι που δεν αρκεί να τους προσκαλέσουν οι υπουργοί για να πιούν ένα καφέ μαζί, αλλά πρέπει να εμπλακούν και αυτοί με τρόπο επικοδομητικό, διότι φέρουν ευθύνη. Τέλος, για τις τροπολογίες όπου εγώ αντιμετωπίζω δυσκολίες τουλάχιστον. Πρώτα, αυτή, αυτό το μίσμα, αυτή η αδυναμία προσαρμογής μεταξύ θέσεων απασχόλησης που είναι κενές και ελλείψεων στις σχετικές δεξιότητες. Πρέπει εδώ πάλι οι επιχειρήσει να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Τέλος, το πρόβλημα της κινητικότητας, επίσης της φυγής των εγκεφάλων. Και τέλος, το πρόβλημα των ανεξάρτητων επαγγελματιών. Αυτά είναι σημαντικά. Έθιξα πολλά βέβαια. Ο δρόμος είναι μακρύς. Έχω όμως την εντύπωση ότι η συνεργασία με τους κοιόδης συζητητές όντως διαμορφώνεται επικοδομητική και πιστεύω ότι θα αποδώσει τις επόμενες εβδομάδες. Ε, Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί την προηγούμενη εβδομάδα όταν έγινε η συνάντηση των σκιωδών δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε ε, γιατί ήμασταν στο Στρασβούργο και δυστυχώς ε, οι υποχρεώσεις ήταν πολλές και πολυπληθείς. Και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε πέρα από τις γενικές σκέψεις που αναφέρθηκαν, το γενικό πλαίσιο, όπως είπε η κυρία Ρέγνερ, ότι δηλαδή θα πρέπει να εντάξουμε αυτή τη συζήτηση στις μακροοικονομικές προοπτικές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανάγκες πέρα από την χειραφέτηση των νέων θα πρέπει να βρούμε οικονομικές οδούς για να τους ενσωματώσουμε στην αγορά εργασίας. Και αυτό δεν το λέω πατερναλιστικά. Ως προς την περιγραφή του θέματος, συμφωνώ με τις προτάσεις. Δεν μιλάμε για συγκεκριμένα μέτρα, αλλά για μία σαφή ανάλυση. Ορισμένες σκέψεις είναι άκρος ενδιαφέρουσες. Ως προς τα δύο βασικά ζητήματα υπάρχουν δύο τροπολογίες που θα θέλαμε να ληφθούν υπόψη. Η μία φορά μία ε, ρήτρα διασφάλισης, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν για την ένταξη των νέων στην αγορά να μην ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελλείμματος, γιατί μιλάμε για ένα συλλογικό μέτρο που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει ευρωπαϊκά. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν του μνημονίου συνεννόησης και στον υπολογισμό του ελλείμματος, αυτές οι ελλείψεις δεν θα πρέπει να υπολογιστούν, να συνυπολογιστούν. Δηλαδή πρόκειται για μία ε, σοβαρή διασφάλιση, για ένα μέτρο διασφάλισης. Να δώσουμε κίνητρα για την εργασία των νέων και για το γενικότερο υπολογισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης ένα πρόγραμμα άμεσης κρούσης έτσι ώστε οι χώρες που έχουν πάνω από 25% ε, ανεργία των νέων να μπορέσουν να δράσουν άμεσα. Έτσι ώστε να απασχοληθούν ένα 10% των νέων που βρίσκονται άνεργοι. Αυτό θα το δούμε και στο Συμβούλιο γιατί ορισμένα κράτη-μέλη ήδη το δέχονται και θα πρέπει να το αναφέρουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως προς άλλες που μας απασχολούν μαζί με την κυρία Ρέγνερ, είναι εκείνες που δημιουργούν σύγχυση μεταξύ αγοράς εργασίας και απασχολησιμότητας των νέων. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτή την αιτιώδη συνάφεια που δημιουργείται πολλές φορές. Γιατί ελοχεύει ένας κίνδυνος και δεν μας βοηθά προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομική βοήθεια των επιχειρήσεων από αυτή την έννοια, γιατί μας ενδιαφέρει η απασχολησιμότητα των νέων. Και δεν ξέρω κατά πόσο η οικονομική διευκόλυνση επιχειρήσεις είναι πάντα το καλύτερο μέσο. Δεν είναι βεβαίως η ίσονος ε, και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τις συμβάσεις σκουπίδια, όπως ονομάζονται, που έχουν σχέση με την ποιότητα της απασχόλησης. Θα πρέπει να έχουμε τα, στα σωστά μέσα, τα κατάλληλα μέσα και να μας ενδιαφέρει η ποιότητα της απασχόλησης καθεαυτής για να καταπολεμήσουμε την επισφάλεια εργασίας που απασχολεί τους νέους. Έχουμε πολλά περιθώρια για να συγκλίνουμε και θα προωθήσουμε τον διάλογο και με τους σκιώδεις για να φτάσουμε σε ένα ευρέως αποδεκτό κείμενο. Ευχαριστώ. Φιλίπ Μπλα, η Νάντια Χίρς και μετά ο συνάδελφος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς την ηγεσία. Ήδη από την πρώτη συνάντηση στο Στρασβούργο τα πήγαμε καλά και βρήκαμε τόπο για να συμβιβαστούμε. Και ελπίζω και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Τα όσα ήδη αναφέρθηκαν με βρίσκουν σύμφωνοι ότι δηλαδή η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων απαιτεί και βραχυπρόθεσμα αλλά και κυρίως μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα βραχυπρόθεσμα βέβαια μέτρα έχουν την έννοια ενός μηνύματος και κυρίως τα χρήματα που είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τρόπο ώστε να προωθήσουμε κάποια μέτρα, να χρηματοδοτήσουμε κάποια μέτρα επιτόπου, να στήσουμε τις πρώτες δομές. Αλλά οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό λέχθηκε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες που επιφέρουν περιορισμό της ε, απασχόλησης των νέων. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε συνεπείς και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, χρειαζόμαστε σαφέστατα διαφορετικές αλλαγές στις διάφορες χώρες. Εγώ θεωρώ ότι η δυτή εκπαίδευση ασφαλώς και είναι καλή, όπως το βλέπουμε και στην Αυστρία και στη Γερμανία, αλλά δεν είναι δυνατόν και να εφαρμοστεί αυτούσια σε όλες τις άλλες χώρες μέλη. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας μέλους. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τις αιτίε της ανεργίας. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τη σχολική εκπαίδευση και εκεί χρειάζονται διαφορετικά μέτρα από ό,τι χρειάζεται κάποιος ο οποίος έχει, για παράδειγμα, το απολυτήριό του, καθώς επίσης και ενδεχομένως και το πτυχίο του Πανεπιστημίου. Εκεί χρειάζεται άλλα μέτρα. Εκεί τη διαφοροποίηση πρέπει να κάνουν οι χώρες μέλη, αναλόγως με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Ίσως μάλιστα να πρέπει να γίνει διαφοροποίηση και στο περιφερειακό επίπεδο των χωρών μελών. Δεν είναι δυνατόν να φαντάζεται κανείς όπως καμιά φορά το μεταφέρουν τα μέσα ενημέρωσης. Α, έχετε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευτυχώς εδώ φανήκαμε πραγματικά πολύ συγκρατημένοι και δεν είπαμε τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τώρα και ορισμένε τροπολογίε δικέ μα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, αυτή την έλλειψη προσαρμογή μεταξύ προσφορά και ζήτηση, αυτό το mismatch. Εγώ δεν το βλέπω τόσο αρνητικά. Ότι δηλαδή με, αυτό, με αυτή τη φυγή κεφάλων μας φεύγουν πάντα οι καλοί. Αν αυτοί οι καλοί δεν βρίσκουν δουλειά, ε τότε έχει καλός. Ας φύγουν οι άνθρωποι αυτοί, ας πάνε σε άλλη χώρα μέλος και ενδεχομένως ορισμένοι να επιστρέψουν, ορισμένοι βέβαια ίσως να βρουν, και κάποιο, εκεί, να βρουν εκεί τον έρωτα της ζωής τους, να πατρευτούν και να μείνουν εκεί. Κάποιοι θα γυρίσουν πίσω όμως στις πατρίδες τους και θα επιστρέψουν και με γνώσεις και δικτυωμένοι και θα δώσουν επομένως τη δυνατότητα μιας ακόμα καλύτερης ανάπτυξης της οικονομίας. Άρα, προς Θεού, μην πούμε «Α, να αποτρέψουμε τον κόσμο να φεύγει από τις χώρες του διότι χάνουμε τους εγκεφάλους». Μιλάμε για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασία. Ίσως μάλιστα αυτή η κινητικότητα να είναι και ένα βήμα για να βγούμε από το τέλος αυτό που αντιμετωπίζουμε. Βρίσκω λοιπόν πολύ λάθος να λέμε ότι κανένας δεν πρέπει να φεύγει από τη χώρα του γιατί έτσι λείπουν εργατικά χέρια ή εγκέφαλοι και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν τροπολογίες οι οποίες τέτοιο περιεχόμενο περίπου έχουν και τις υποστηρίζουμε αυτές. Το ίδιο για τον ανεξάρτητο επαγγελματία. Πού αξίζει τον κόπο να ληφθεί υπόψη. Ασφαλώς. Να μην είναι ψεύδο ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, που μετά από ένα εξάμεινο να πτωχεύσουν, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους που καμιά φορά έχουν πολύ καλές ιδέες και σε όλη αυτή την υπόθεση του διαδικτύου κτλ. Και, και οι οποίοι γνωρίζουν και πώς λειτουργεί το διαδικτύο. Αυτοί πρέπει να κινητοποιηθούν και να τους προσφέρουμε κίνητρα δηλαδή. Τέλος, ο υπολογισμός του ελλείμματος. Ασφαλώς, μέτρα στον τομέα της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να αφαιρούνται από το έλλειμμα. Τότε φοβούμε ότι όλα θα βαφτιστούν μέτρο απασχόλησης των νέων, μπορεί να είναι και μέτρα τα οποία δεν είναι διόλα αποτελεσματικά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές. Να πούμε δηλαδή ότι δεν μπορούν να μπουν εκεί μέσα όλα τα πράγματα αυτά γιατί τότε μπορεί να προκύψει κατάχρηση από τις διάφορες χώρες μέλη. Όπως είπα, να δηλωθούν όλα όσοι δίθεν μέτρα για την πρόθεση της απασχόλησης των νέων. Τα χρήματα που θα δοθούν πρέπει να ταπανηθούν και πραγματικά αποδοτικά. Έχουμε λοιπόν πολλές τροπολογίες που ευχαρίστως εμείς θα αναζητήσουμε συμβιβαστικέ τροπολογίες στην βάση τους και έτσι στη βάση αυτή να συνταχθεί η έκθεση. Φιλιππουλά. Ε, είναι, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Έχει κατεπίγοντα χαρακτήρα. Και αυτό είπε και η κυρία Ρέγνερ, ε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ε, σε αυτή την κατεπίγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι, αυτή την, ε, αυτό τον όλεθρο, αυτή την καταστροφή. Άρα δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που προελέχθησαν. Ε, απλώς ε, να πω τι ανακύπτει και από τις τροπολογίες θα πρέπει να απλουστεύσουμε το, τα διοικητικά διαβήματα έτσι ώστε ε, να υπάρχουν ενίες θηρίδες πρόσβασης και διαρθρώσεις που να μας επιτρέψουν ε, να προωθούμε τους νέους σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα από μία ενιαία θηρίδα ε, με βάση τη, τις κοινωνικές ε, συνιστώσεις, ιατρικές και ούτω καθεξής για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους και να τους ε, διευκολύνουμε στο να έχουν μια άδεια οδήγησης, πρόσβαση στο σύστημα υγείας, κατάρτιση και να βοηθήσουν και τα κρατη πέρα από τις ε, κλασικές διαρθρώσεις απασχόλησης και απασχολησιμότητας, δηλαδή τέλειο τους καταλόγους θέσεων για τους νέους. Θα ήθελα να δώσουμε δυνατότητα στους νέους μέσω εθελοντισμού, ε, πληρωμένης μαθητείας έτσι ώστε ε, όλα αυτά να συνυπολογίζονται ως ε, επαγγελματική εμπειρία και να μην θεωρήσουμε ότι οι ναι, νέοι δεν έχουν πείρα γιατί δεν έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου, για παράδειγμα. Δηλαδή να αξιολογούμε και αυτές τις περιόδους μαθητείας για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού τους. Και επίσης η κατάρτιση, να δούμε την κατάρτιση και τις εναλλασσόμενες περιόδους μαθητείας. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη μικροχρηματοδότηση, στα επιμέρους προγράμματα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους ιδιώτες αν θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους ε, δηλαδή επιχείρηση. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερα στη χώρα μου. Και τα 6 δις ευρώ για την επόμενη επταετία αποτελούν αμεληταίο ποσό αν δούμε ποιο είναι το διακύβευμα, δηλαδή τη βοήθεια των νέων ε, για να απασχοληθούν. Επίσης ε, θα πρέπει να διεισδύσουμε στο σχολικό, στον κόσμο του σχολείου για να μην εγκαταλείπουν οι νέοι το σχολείο. Ε, εγώ από όσο γνωρίζω ε, ήδη από το σχολείο δεν προωθούνται ορισμένες διαρθρώσεις, δηλαδή δεν βλέπουμε τις πραγματικές ανάγκες ε, ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Άρα πολλοί εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί δεν τους ε, προσανατολίζουμε, τους κατευθύνουμε προς τις πραγματικές ανάγκες. Πρόκειται για τους νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και δεν έχουν ε, την δυνατότητα ούτε κοινωνικά ούτε διανοητικά να κινηθούν τάχιστα, να έχουν τη σωστή κατάρτιση και όλα αυτά κοντά στην κατοικία τους και στην οικογένειά τους για να γίνουν και οι κατάλληλες εξοικονομήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να διεισδύσουμε στο σχολείο για να υπάρξει ε, διασυνδεσιμότητα μεταξύ του σχολείου και του επαγγελματικού κόσμου πολύ κοντά στα σχολεία. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ε, νέους να μην εγκαταλείψουν το σχολείο και να έχουν πρόσβαση και στον κόσμο της εργασίας. <coughs> ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, αλλά όταν ε, παρουσιάσατε την έκθεσή σας, όταν αποφασίσαμε για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και την εξετάσαμε, δυστυχώς ε, μας ε, κατέλαβαν τα γεγονότα, μας προσπέρασαν μάλλον και αυτό το λέω δυστυχώς γιατί έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και οι πρωτοβουλίες πολλαπλασιάζονται. Έχουμε και την ανακοίνωση του Επιτρόπου Άντορ, τη σημερινή ανακοίνωση που ενέκρινε σήμερα το Διευθυντήριο για την απασχόληση των νέων και που επαναλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες που ήδη γνωρίζουμε σε αυτόν τον τομέα. όπως ε, αναμένεται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε τις προτάσεις που είχαμε και δεν προβάλλουν κάτι νέο από πλευράς του πολιτικού κόσμου, του πολιτικού στερεώματος. Η έκθεση πρωτοβουλίας αφορά ένα ευρύτατο θέμα. Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα που έχει κινητοποιήσει πολλούς. Μιλάμε για 331 τροπολογίες, αλλά θα πρέπει να στοχοθετήσουμε καλύτερα τα 3-4 βασικά μηνύματα, τα οποία να είναι πιο ε, πρωτότυπα από αυτά που διαβάζουμε στα συνήθη συμπεράσματα και να αποτελέσουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Τέλος, σε αυτά που είπατε για έναν αξιοπρεπή μισθό, παρακολουθώντας εργασίες του ΩΣΑ, τις οποίες απηχούσαμε και εμείς, απηχούμε και εμείς αφορούν μία αξιοπρεπή, την αξιοπρεπή εργασία, έναν αξιοπρεπή ε, μισθό. Και αυτό το βλέπουμε και στις ε, διάφορες διακυβερνητικές, στις μη κυβερνητικές που μας μίλησαν στην πρόθεση αυτής της έννοιας του αξιοπρεπούς μισθού διότι με την κρίση έχουμε τους ε, λεγόμενους φτωχούς ε, μισθωτούς ή εργαζόμενους. Γι' αυτό αποτελεί μια βασική έννοια, θα πρέπει να το δούμε και στις περιόδους και για τις περιόδους μαθητείας. Πώς θα προωθήσει η Επιτροπή ένα πλαίσιο για τους μαθητευόμενους αυτό το είδαμε στην έκθεση του Ρίνεν, καθώς και την πλαισίωση των περιόδων μαθητείας, για να μην υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε μαθητευόμενος θα πρέπει να αμείβεται με τον ελάχιστο μισθό, αλλά με έναν αξιοπρεπή τουλάχιστον. να υπάρχει μία ανταμοιβή, αν δεν θέλετε να μιλήσουμε για μισθό. Δεν μπορούμε να το λύσουμε ολοκληρωτικά. Υπάρχουν οι περίοδοι μαθητείας που οργανώνονται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση. όταν μιλάμε εκτός επαγγελματικής κατάρτισης για άλλες, ε, άλλου τύπου μαθητίας, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για αξιοπρεπή μισθό. Ε, γιατί διαφορετικά μιλάμε για νέες μορφές εκμετάλλευσης των νέων. Η Επιτροπή δεν θέλει το λόγο, δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καταρχήν θα ήθελα να απαντήσω στις δικές σας παρεμβάσεις. Πράγματι, όσον αφορά τις ε, πρωτοβουλίες για τους ε, νέους, έχουμε όλο ένα και περισσότερες. Και η απόδειξη είναι ότι δεν, είναι ποτέ, δεν επαρκούν ποτέ. Ε, στην έκθεσή μου στην έκθεση μου προσπάθησα να διατυπώσω μακροχρόνιες λύσεις, τις βέλτιστες δυνατές για την αγορά εργασίας των νέων και να δείξω, να καταδείξω τα προβλήματα ε, σε διάφορα επίπεδα. διότι όλοι συμμετέχονται στα κράτη-μέλη η περιφερειακή θεσμοί, όπως είπε και η κυρία Χίρς, δεν επαρκούν. Όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Δεν μπορούμε να εκμηδενήσουμε την ανεργία αυτή, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον θα μειωθεί η ανεργία σύντομα. Στην Ελλάδα, η οποία πλήττεται ιδιαίτερα, συμβαίνει το ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει μία παλινοδία της κατάστασης. Θα πρέπει να δούμε ε, πώς ε, η Ελλάδα και οι χώρες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το θέμα, φάνοντας και σε έναν αξιοπρεπή μισθό, δηλαδή ένας μισθός που να αντικατοπτρίζει την ε, παρεχόμενη εργασία. Οι περίοδοι μαθητείας θα πρέπει να αμείβονται. Αυτό το είδαμε και στα πλαίσια της ε, ε, πρότασης της κυρίας Φοντένα. Θα πρέπει να αμείβονται οι μαθητευόμενοι και θα πρέπει να τονίσουμε ότι και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε πάντα έντιμοι γιατί δεν δίνουμε πάντα, δεν αμείβουμε πάντα σωστά το βοηθητικό μας προσωπικό θα πρέπει να δούμε πώς ορίζεται ο μισθός του βοηθού, πώς ακριβώς προσδιορίζεται, πώς ε, καταβάλλονται οι δαπάνες ε, ε, μετάβασης ταξιδιού, γιατί η μαθητεία δεν σημαίνει εκμετάλλευση των νέων και συμφωνώ μαζί σας, γιατί εάν η μαθητεία υπερβεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά δηλαδή τους 12 μήνες, τότε θα πρέπει να μετατρέπεται σε σύμβαση εργασίας, γιατί όποιος έχει εργαστεί 12 μήνες έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη εμπειρία. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι μισθωτός. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα ημέτερα. Ας βάλουμε τάξη στα ημέτερα πριν ε, το απαιτούμε από τους άλλους. Σε σχέση τώρα με τον υπολογισμό του ελίματος, ε, συμφωνώ με τη θέση της Νάντια Χίρς. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι δεν γίνονται κατάλληλε ε, δαπάνε στα κράτη-μέλη. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, το προηγούμενο μήνα ο Υπουργός Εργασίας κατάρτισε τα προγράμματα για τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας. Ελπίζω να καταλήξουν κάπου ως προς τους αυτοαπασχολούμενους. Θα λάβω υπόψη της υποδείξεις των σκιωδών. Πρόκειται για επισφαλή εργασία πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε και τη, τους αυτοαπασχολούμενους μέσα στα πλαίσια της ε, επιχειρηματικότητας. Δεν θέλουν όλοι να είναι μισθωτοί υπάρχουν ε, άνθρωποι που προτιμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να δράσουν ε, αυτόματα, να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Θα ήθελα λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την ε, συλλογιστική που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή από όλους. σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα μεταξύ σχολείου και αγοράς εργασίας, να υπάρχει μια ρευστότητα και μια προσαρμογή ανάλογα με τα προσόντα και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μίλησα για τη σημασία που θα πρέπει να δώσουμε ε, στο σχολείο και νομίζω ότι θα πρέπει να δράσουμε και σε περιφερειακό επίπεδο, διότι πολλές φορές οι νέοι που να αποφασίζουν για τη σταδιοδρομία τους δεν έχουν σαφή ιδέα για το τι θα κάνουν στο μέλλον, σε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν εργασία και που θα είναι πιο εύκολο να βρουν αυτή τη θέση εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει βοήθεια από τα περιφερειακά συμβούλια για να βοηθήσουμε τα παιδιά στη σταδιοδρομία τους, εκεί όπου υπάρχουν ε, περισσότερες θέσεις εργασίας. Με συγχωρείτε, ξέρω ότι θα γίνουν και άλλες συναντήσεις με τους σκιώδεις και ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα ζητήματα, να φτάσουμε σε λύσεις που θα μας επιτρέψουν να σας ικανοποιήσουμε, ελπίζοντας ότι θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση των νέων αγοριών και κοριτσιών Α, ξέχασα ως προς την κινητικότητα. Το είπα δύο φορές στην παρουσίαση της έκθεσης. Δεν είμαι και τόσο υπέρμαχη της ε, ιδέας αυτής ότι θα πρέπει κανείς να εγκαταλείψει τη χώρα του για να βρει εργασία θα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Δηλαδή τι προτιμούν τα παιδιά να παραμείνουν στη χώρα τους ή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ισχύει η αρχή του το μη βέλτιστον, δηλαδή να βρει κανείς ε, εργασία και εκτός της χώρας του. Ε, πάνω από ένα εκατομμύριο νέων Πολωνών ζουν ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και δεν είναι όλοι νέοι. Ένα εκατομμύριο βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και αλλού γιατί δεν μπορούν να βρουν θέση εργασίας στη χώρα τους. Η κατάσταση αλλάζει άρδιν και θα πρέπει να αποφασίσουν πολλοί νέοι δυστυχώς να εγκαταλείψουν την χώρα τους. Πολλοί είναι εκείνοι λοιπόν που πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα τους, αλλά πολλοί επιστρέφουν και χρησιμοποιούν ε, τις γνώσεις αυτές στην ε, Πολωνία και έτσι η Πολωνία κερδίζει πολλά από αυτούς ε, τους νέους που επιστρέφουν στη χώρα τους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για τις παρατηρήσεις σας. Ελπίζω η εργασία να είναι ικανή. Euh, Ευχαριστούμε και σας εύχομαι κουράγιο για την ε, εκπόνηση των συμβαστικών τροπολογιών που θα συζητήσουμε στις 8 Ιουλίου. Και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το απόγευμα. Πρόκειται για την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας επί της έκθεσης του κ. Προύστ για την Επιτροπή Ήτρε και πρόκειται για την πρωτοβουλία CARS 2020. Είναι ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Το λόγο έχει η συγγητριά μας, η κυρία Birgit Σίπελ, για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ιδίως ευχαριστώ που επιτρέψατε να βάλουμε προς το τέλος της συνεδριάσεως το θέμα ώστε να μπορέσω να σας παρουσιάσω εγώ ίδια την ε, γνωμοδότησή μου. Χάρηκα για την πρωτοβουλία της Κομισιόν διότι καθιστά σαφές και ιδίως εν μέση οικονομική κρίση ότι παρόλη τη σημασία του τομέα των υπηρεσιών Παρ' όλα αυτά είναι απαραίτητη μια στέρεα βιομηχανική βάση για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτών. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας παίζει βέβαια ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο με, με 12.000, 12 εκατομμύρια φυσικά, 12 εκατομμύρια εργαζόμενους και στις αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά βέβαια και στις πολλές εταιρείες που προμηθεύουν εξαρτήματα κτλ. Εκεί άλλωστε γίνονται και οι περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και σε καινοτομία και σε έρευνα. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού αυτού τομέα, αλλά και για την διατήρηση της πρωτοπορίας μέσω των επενδύσεων και βέβαια της βιωσιμότητας της απασχόλησης που για μας εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης παίζει κέριο ρόλο. Γι' αυτό στη γνωμοδότησή μας αναφερόμαστε έμεσα βέβαια μόνο στις μελλοντικέ προοπτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας, κυρίως όμως ασχολούμαστε με την κατάσταση των απασχολούμενων και με τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον τομέα αυτό ο οποίος και διαρκώς αναπτύσσεται. Γνωρίζουμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ιδιαίτερα δυναμική αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, το βάρος των αυτοκινήτων οχημάτων, όπου πολλά πράγματα αλλάζουν και γι' αυτό επέρχονται πολλές αναδιαρθρώσεις που βεβαίω δεν είναι δυνατόν να απευθυνθούν. Μέσα στα πλαίσια αυτών των αναδιαρθρώσεων οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι πρέπει να διαβουλεύονται με τους άλλους φορείς και οι εμπειρίες του παρελθόντος δείχνουν ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν θετική απήχηση και θετικό αποτέλεσμα. Ε, επιτρέπουν και την περαιτέρω χρήση των εμπειριών των εργαζομένων. Και επειδή η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι μονάχα επιτυχημένη, είναι όμως και πολύ στενά δικτυωμένη με στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν σκόπιμο εάν για τις αναδιαρθρώσεις αυτές στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ελάχιστες προδιαγραφές, έτσι ώστε να γίνει αυτό ευκαιρία όχι μόνο για τον κλάδο, αλλά για τους βιομηχάνους δηλαδή, αλλά και ιδίως για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους. Εν προκειμένου παίζει ιδιαίτερο ρόλο και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, το οποίο έχει σαφώς θετικές επιπτώσεις. Πιστεύω δε ότι οι χώρες μέλη στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα κατορθώσουν να βρουν λύση τις ημέρες αυτές που είναι εποφελής για όλες και όλους. Είπα ήδη ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ιδιαίτερα εύκαμπτος, ευέλικτος, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικές, σημαντική και η ανάπτυξη των προσόντων των εργαζόμενων. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν της δημιουργίας δηλαδή ενώ συμβουλίου της κατάρτισης των εργαζόμενων στις αυτοκινητοβιομηχανίες για να δούμε ποιες είναι οι γνώσεις που απαιτείται να διαθέτουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις σχετικές προκλήσεις και ιδίω βέβαια μέσα στα πλαίσια μιας διαρκούς κατάρτισης που έχει ιδιαίτερη σημασία. Εκεί βέβαια καλούνται και οι χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές και να τις εντάξουν μέσα στα, στους μελλοντικούς τους σχεδιασμούς, να λάβουν δε τα απαραίτητα μέτρα. Ακούσαμε ήδη τα σχετικά περί κινητικότητας, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί με διαφόρους τρόπους και που είναι σημαντικό εν προκειμένου ανεξαρτήτως τώρα της απόψεως που έχουμε για την κινητικότητα αν την κρίνουμε θετικά ή λιγότερο θετικά για τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες είναι σημαντικό να είναι ενήμερες και ενήμεροι για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά των και διαμεθοριακά και να μπορούν να μετακινούνται και να διακινούνται με την απαραίτητη ασφάλεια χωρίς να υπάγονται σε κινδύνους για, την, για τον ε, σχεδιασμό του βίου τους. Βεβαίως η γνωμοδότηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί κάποια στενά όρια θα έλεγα όπως γνωρίζετε, συντομία δηλαδή. Γι' αυτό αναμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων, επί των οποίων θα συζητήσουμε, ώστε να βάλουμε κάπως περισσότερη σάρκα στον σκελετό που παρουσιάζω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση αυτή για την Επιτροπή μας, αλλά και για το μέλλον της αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Και δεν ισχύουν αυτά μόνο για αυτόν τον οικονομικό κλάδο, αλλά και για πολλούς άλλους. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η συγγήτρια παρόλο που είχε λίγο χρόνο για να ετοιμάσει την έκθεσή της, το φρόντισε, περιλαμβάνουν τα σημαντικά σημεία. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των αυτοκινήτων που φτιάχνουμε. Αυτό θα μας διαφοροποιήσει σε σχέση με άλλες αγορές. Αν λοιπόν επενδύσουμε σε προηγμένη τεχνολογία, όπως είπε και η συγκήτρια, και αν στοιχηματίσουμε στην καινοτομία, τότε θα μπορέσουμε και να πετύχουμε. Οι εργαζόμενοι επίσης στον κλάδο πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο για να αλλάξουν οι εργαζόμενοι, να αποκτήσουν δηλαδή τα προσόντα που χρειάζονται για να απασχοληθούν σε αυτό το τομέα. Να γίνει αυτή η μετατροπή. Όταν λέμε ότι πρέπει να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από την άλλη ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τα πάντα. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε εδώ τους εργαζόμενους να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ορίζοντας 2020 το πρόγραμμα COSME που μπορούν να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να υποφεληθούν έτσι. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το θέμα της αναδιάρθρωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Στην έκθεση Θέρκας λέγαμε ότι πρέπει να προλάβουμε τις καταστάσεις. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Από τη δικιά μου περιφέρεια. Αραγών. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη, πιο μεγάλη επιχείρηση που είναι General Motors. Μια από τις πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως γενικά υπήρχαν προβλήματα, έτσι υπήρχαν και εκεί, κατάφερε όμως να πετύχει συμφωνία η επιχείρηση με τους εργαζόμενους εκεί, τα συνδικάτα. Τι πέτυχαν προλαμβάνοντας τις καταστάσεις, την αναδιάρθρωση να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης, να τηρούνται οι παύσεις, η νυχτερινή βάρδια που πήγαινε να καταργηθεί, πάγωμα των μισθών για φέτος και του χρόνου και κάποιες μικρές περικοπές. Έτσι όμως δεν χάθηκε καμία θέση απασχόλησης. Να λοιπόν ένα καλό παράδειγμα που προλαμβάνει την αναδιάρθρωση. Ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία με την εισηγήτρια να μιλήσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στις εργασίες που έγιναν στα πλαίσια της έκθεσης Σάρκας και εσείς το αναφέρατε επίσης κυρία Λόπε Φοντανιέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που την έχουμε εδώ και ένα μήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν έχει αντιδράσει. Θα θέλαμε να έχουμε ένα δελτίο πληροφοριών στο οποίο να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα κάνει διαβουλεύσεις αλλά όχι μόνο αυτό γιατί αυτό δεν φτάνει όταν πρόκειται για μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Ίσως και εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση Κριτσπέρκ για να επενθυμίσουμε τι ψηφίσαμε στα πλαίσια της έκθεσης Θέρκας. Η απάντηση της Επιτροπής δεν μας ικανοποιεί μέχρι τώρα. Ενώ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας η αναδιάρθρωση είναι πολύ σημαντική και εφόσον γίνεται καλά είναι κάτι θετικό. Η συγκήτρια τώρα έχει το λόγο για να απαντήσει ίσως την κυρία Λόπε Φωτανιέρ και έτσι θα ολοκληρώσουμε και τις εργασίες μας. Παρακαλώ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη αφού ευχαριστήσω πρώτα για τις, ε, για τις παρατηρήσεις σας Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα όντως, ευχαριστώ για τη σχετική παρατήρηση, ειδικά για το θέμα των αναδιαρθρώσεων, να το τονίσουμε δηλαδή ιδιαίτερος και την αξία για την βιομηχανία, για τους εργαζόμενους να ασκήσουμε δε ταυτόχρονα κάποια πίεση. Για το θέμα της εκπαίδευσης για μένα είναι σημαντικό να δεχθεί ότι ιδίω στην αυτοκινητοβιομηχανία γίνεται πολύ υπεραιτέρω κατάρτιση και ανεξάρτητα μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις και μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα και να χρηματοδοτηθούν από τις ίδιες. Βεβαίω πάντοτε μπορούν να μπουν κάποιες συνθήκες πλαίσια γιατί είναι σημαντικό να γίνει υπεραιτέρω κατάρτιση ιδίω για τους νέους ε, συνεργάτες. Και αυτά τα πράγματα να γίνουν πανευρωπαϊκά, ώστε να αποκτώνται αυτά τα προσόντα. Ευχαριστώ τη συνάδελφο, διότι εκτός από την αυτοκινητοβιομηχανία και τους προμηθευτές της, τόνισε ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς της βιομηχανίας οι οποίοι θίγονται και δεν μπορούν να μείνουν εκτός παρενθέσεως. Χαίρομαι λοιπόν πράγματι για τις παραπέρα συζητήσεις που θα κάνουμε και πιστεύω και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια έκθεση που βεβαίως θα έχει ένα πλουσιότερο περιεχόμενο από ό,τι είναι δυνατόν να γίνει στο σχέδιο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών 2 Εβδόμου. Εξετάζουμε το κείμενό σας 5 Ενάτου. Εξετάζονται οι τροπολογίες στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 26 η ψηφοφορία. Και η Επιτροπή Ήτρε θα ψηφίσει την έκθεση επί της ουσίας στις 18 Δεκάτου. Εδώ λήγουν οι εργασίες για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 9 και 10 όπου βέβαια θα είναι η συνεδρίαση αφιερωμένη μοναχά στις ψηφοφορίες. Οπλιστείτε με τις κάρτες σας και υπομονή.